συγχρόνων υπηρεσιών κινητών δεδομένων. Καλύτερα από ό,τι στην ΗΠΑ και στην Κίνα. Αλλά απαιτεί αυτό να ασκήσουμε πίεση συνεχή και τα επόμενα χρόνια γιατί δεν είμαστε έτοιμοι αλλά οι αποφάσεις που λαμβάνουμε τώρα δίνουν στην ευρωπαϊκή βιομηχανία συνολικά γιατί το θέμα δεν αφορά μόνο τις λεπικοινωνίες αφορά τη βιομηχανία και την οικονομία τις καλύτερες προϋποθέσεις και ε, να έχουμε ένα αρκετά μεγάλο απόθεμα θα έλεγα όσον αφορά τις συχνότητες για το μέλλον. Νομίζω επίσης πως τα καταφέραμε όσον αφορά την αυστηρότητα των κανόνων ανταγωνισμού και επιτύχαμε περισσότερα από ό,τι σε άλλους τομείς, αλλά ε, Τώρα, ε, στο τέλος των διαπραγματεύσεων, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις ομάδες και ιδιαίτερα τον κύριο Ρόιλο, ο οποίος προείδρευσε στον ε, τριμερή διάλογο. Όπως και στην Επιτροπή μας, είναι πρόεδρος αυστηρός που επιτυχάνει αποτελέσματα. Ελπίζω λοιπόν να στηρίξετε τη συμφωνία αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Περνάμε στην ψηφοφορία, ηλεκτρονική ψηφοφορία, γιατί είναι το σύνολο του κειμένου, άρχιτη ψηφοφορία. doesn't work. Δεν δουλεύει, μια στιγμούλα, μια στιγμούλα. Der, du musst mal, der Johansson, der hat seine Karte. Yeah, Να περιμένουμε λίγο. Εντάξει, πέρας. Ωραιότατα, συγχαρητήρια κύριε Χέκμαρκ. Ε, νομίζω θετικά τα πράγματα, συνάδελφοι. Έχετε πρόβλημα με την κάρτα? Ah, συν, συν δύο ακόμα. Τρεις ακόμα. Τρεις μηχα... Τρία μηχανήματα δεν δουλεύουν. Ακόμη μεγαλύτερη λοιπόν η πλειοψηφία. Μετά πρέπει να ψηφίσουμε την επιστολή που πρέπει να απευθύνουμε στην Πολωνική Προεδρία. Ποιο είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. Περνάμε σε επίθεση των πληροφοριακών συστημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έχετε τα έγγραφα. Μια στιγμούλα. Ξεκινάμε. Ναι με την 41. 41 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 42 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 43 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 44 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 45 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 46 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 8 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 9 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 50 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Περνάμε. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 11 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 55 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 6 κατά αποχές δεκτή 30 υπέρ κατά αποχές δεκτή 31 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 36 υπέρ κατά αποχές δεκτή 37 υπέρ κατά αποχές δεκτή 38 υπέρ κατά αποχές δεκτή 39 υπέρ κατά αποχές δεκτή 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή 40 υπέρ κατά Αποχές. Δεκτή. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική. Άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρας. Σαράντα υπέρ, μία αποχή. Λειτουργήσαν όλες οι συσκευές, ωραία. Όχι. Όλα εντάξει. Έλερ. Δύο φράσεις να πω. Μιλούμε για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Για, πρώτη φορά εξετάσαμε το νομικό πλαίσιο στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι σε όλα τα κράτη-μέλη πέρσι 32 υποθέσεις εγκλήματος του κυβερνοχώρου πήγαν στα δικαστήρια και μόνο 11 κατέληξαν σε καταδίκη. Και για πρώτη φορά έγινε προσπάθεια συντονισμού σε ρυθμιστικό επίπεδο για να συντονιστούν οι προσπάθειες στα κράτη-μέλη. Δεύτερον, ευχαριστώ που περιορίσαμε το πεδίο της έκθεσης στην νομοθεσία της Επιτροπής, διότι η καθήλια αρμόδια Επιτροπή απεφάσισε ότι θα λάβει υπόψη όλες τις τροπολογίες μας στην έκθεσή τους. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος όχι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον συντάκτη, τον κύριο Έλερ. Περνάμε σημείο 6. Οικονομική κρίση στον αμυντικό τομέα. Ο κύριος Τζενόφσκι το προετοίμασε. Περνάμε στις ψηφοφορίες. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική όχι. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15 σε 2 μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική τρία υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρι... Εγκρίνεται με συγχωρείτε. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 30 υπέρ με προφορική τροπολογία υπέρ κατά να ξαναδώ ποιοι είναι υπέρ ευχαριστώ ωραία κατά εντάξει δεκτή 32 υπέρ 32 υπέρ καταπίπτει 29 γράφει εδώ πέρα Καταπληκτή, Ναι. Ωραία. 32 υπέρ. Κατά. Υπόλοιποι. Υπέρ. Ωραία. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 37 υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Οπότε περνάμε 44 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 45 υπέρ. Κατά. Ποιοι είναι υπέρ τη 45 ξανά. Να επαληθεύσουμε. Ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Και περνάμε στο σύνολο της έκθεσης, ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Και δεκτή συγχαρητήρια κύριε Τόζενόφσκι. Περνάμε άρα στο σημείο 7 αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 και εδώ πέρα υπάρχει ένας κατάλογος συναδέλφου Σαρτόρη τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 4 υπέρ. 6 με συγχωρείτε υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 10 υπέρ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 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή 32 υπέρ ε, 23 με συγχωρείτε υπέρ κατά αποχές δεκτή 24 υπέρ συγγνώμη κυρία Τικάου Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω ότι αναφερόμαστε στις μελλοντικέ ανάγκες χρηματοδοτήσεως του ΙΤΕΡ. Θα ήθελα, συνεπώς, να έχουμε την γνωμοδότηση της Επιτροπής πριν ψηφίσουμε την τροπολογία αυτή για την ανάγκη αναλύσεως επί των μελλοντικών χρηματοδοτήσεων ΙΤΕΡ, βάσει των project bonds θα ήθελα την άποψη της Επιτροπής πριν ε, να ψηφίσω. θα το δούμε πριν την, ε, τελική ψηφοφορία, εντάξει, ίσως να είναι λίγο ασύνηθες. Όχι, συνήθως ψηφίζουμε. Αν υπάρχει κάποια αντίρρηση θα, θα τηρήσω τον κανόνα. Λοιπόν, 23 ήταν το επόμενο, υπέρ. Το ψηφίσαμε κιόλα. Α, συγγνώμη, 24. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Περνάμε λοιπόν στην τελική ψηφοφορία. Ε, με ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται. Πέρα. Και γίνεται δεκτή συγχαρητήρια στην εισηγήτρια τελείωσε αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Τελείωσαν οι ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ζητώ κατανόηση, έπρεπε να τηρήσω τους κανόνες. Θα ήθελα να συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες συζητήσεις, αλλά λίγη ησυχία στην αίθουσα. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ, οι συζητήσεις εκτός της αίθουσας, έτσι ώστε όσοι θέλουν να συνεχίσουν να μην χρειάζεται να φωνάζουν. Ε, μα δεν είναι δυνατόν. Συνάδελφοι, Συζητήσεις εκτός της αιθούσης, παρακαλώ. Για να συνεχίσουμε εμείς εδώ πέρα. Not always. Sometimes the thing refuses. Gibt es hier so ein Bing-Bang? Und Geräusche? Ξεκινάμε. Περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα αναδιατύπωση. Τον λόγο θα λάβει αποκλειστικά η κυρία Νίμπλερ. Η υπόλοιπη σημαίνει ότι δεν θα μιλάνε άρα. Καλό είναι να την ακούσετε κιόλα. Κυρία Νίμπλερ, έχετε το λόγο εσεί και μόνο. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα διεξάγεται η πρώτη συζήτηση για, με βάση τη νέα πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον κανονισμό για την περιαγωγή υπαριθμών 3. Θα ήθελα να κάνω μια εισαγωγή στο θέμα και θα ήθελα να ακούσω και τι απόψει όλων σα, να έχω κάποιε πληροφορίε από εσά πριν αναφερθώ στην ουσία τη προτάσεω τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πριν σας δώσω τις πρώτες μου εντυπώσεις, την πρώτη μου αξιολόγηση, θα ήθελα να κάνω κάποια πρώτα σχόλια. Ξέρετε ότι συζητούμε το θέμα του roaming της περιαγωγής επί σειρά ετών στο Κοινοβούλιο. Το 2007 υιοθετήσαμε τον κανονισμό roaming 1 και για πρώτη φορά ετέθησαν οροφές στις τιμές για τηλεφωνήματα εισερχόμενα και εξερχόμενα επικινητών τηλεφώνων. Το 2009 θεσπίσαμε τον κανονισμό Roaming 2 που αφορούσε και τα μηνύματα SMS και τη μεταφορά δεδομένων. Και γενικότερα θεσπίσαμε τις υπηρεσίες. Από τον Ιούλιο οι πελάτες της περιαγωγής του roaming ξοδεύουν στο μέγιστο 39 ευρώ για εξερχόμενα τηλεφωνήματα και 15 για εξερχόμενα τηλεφωνήματα. Και τα SMS δεν θα έπρεπε να κοστίζουν πάνω από 11 ευρώ το μήνα. Και όσον αφορά και τα, την περιαγωγή στοιχείων, data roaming, η οροφή είναι 80 ευρώ. Αυτό αποφασίσαμε το 2007. Γιατί? Διότι είδαμε ότι υπάρχουν υπερβολικές τιμές που εφαρμοζόταν και στα 27 κράτη-μέλη και αν κάποιος τηλεφωνούσε διασυνοριακά ή αν έστρανε SMS ή αν κατέβαζε στοιχεία στο τηλέφωνό του, κόστισε μια περιουσία. Αυτό ήταν γελίο σε μια εσωτερική αγορά. Έχουμε εσωτερική αγορά επί έτη για τις τηλεπικοινωνίες, οπότε η κατάσταση ήταν εντελώς γέλια. Ποια είναι η κατάσταση τώρα. Πρέπει να σας πω ότι η κατάσταση βελτιώθηκε κάπως όσον αφορά τους κανονισμούς 1 και 2 για την περιαγωγή και τα εισερχόμενα τηλεφωνήματα κοστίζουν 46% λιγότερο πριν εφαρμοστεί η νομοθεσία για την περιαγωγή. Όμως υπάρχουν φοβερέ τιμέ ακόμα που πληρώνονται για τη μεταφορά δεδομένων. Είναι πολύ ψηλέ για μεταφορά δεδομένων σε περιαγωγή. Και είναι καλό που έκανε την πρόταση ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περιαγωγή 3, roaming 3, για να είναι πιο φιλικέ οι τιμέ για τον καταναλωτή όσον αφορά και τα στοιχεία, τα δεδομένα. Αυτή είναι η βάση τη προτάσεω και, και όλοι ξέρετε ότι το επόμενο καλοκαίρι οι κανονισμοί roaming 1 και 2 θα εκπνεύσουν. Και γι' αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε να, να παραμείνουν οι τιμές και μετά το επόμενο καλοκαίρι καλές τιμές για τους καταναλωτές. Και γι' αυτό πρέπει να κινηθούμε γρήγορα εμείς για να ετοιμάσουμε τον κανονισμό για την περιαγωγή παριθμών 3, roaming 3, για να μην υπάρχει νομοθετικό κενό. Θέλουμε ο νέος κανονισμός roaming 3 να τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την εκπνοή των άλλων δύο. Τώρα, όσον αφορά την ουσία της Ποτάς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπάρχει κάποιο καινοτόμο στοιχείο Υιοθετήσαμε τον κανονισμό για την περιαγωγή όχι διότι θεωρούσαμε ότι ήταν άριστη λύση οι οροφήσει τιμέ στην Ευρώπη. Όχι, ο στόχο ήταν να έχουν περισσότερο ανταγωνισμό στην αγορά. Αυτό ήταν ο βασικό στόχο. Και σύμφωνα με την ανάλυση των τελευταίων ετών, ε, είδαμε ότι δεν το έχουμε πετύχει αυτό. Δεν καταφέραμε να φέρουμε περισσότερο ανταγωνισμό στην αγορά των τηλεπικοινωνιών. Γι' αυτό καλωσορίζω την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλουμε να συνεχίσουμε απλώς βάση ανωτά των ορίων στις τιμές, όχι μόνο βάση αυτού, αλλά θέλουμε να υπάρχουν και ανώτατα όρια στην περιεγωγή, στην τελική τιμή πληρώνει ο καταναλωτής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει διαθροτικά μέτρα στην πρότασή της για αυτό το σκοπό. Ότως ώστε οι εξερχόμενες εταιρείε να διευκολυνθούν να γίνει, να γίνει απεμπλοκή, να υπάρξει unbundling, απεμπλοκή των ε, δικτύων για να βοηθηθούν. Ε, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε στη ρίζα το πρόβλημα, σωστά το θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να μπορέσουμε να εγγυηθούμε ότι υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός στην αγορά αυτή. Ε, στόχος μας είναι να έχουμε εσωτερική αγορά στον τομέα που να λειτουργεί. Ε, δεν θέλουμε απλώς μια ξερή αριθμιστική προσέγγιση που θα θέτει οροφές για τα επόμενα 10-15 χρόνια. Θέλουμε να πιεστούν προς τα κάτω τα ανώτατα όρια, οι οροφές και όσον αφορά τα προτινόμενα ανώτατα όρια για, για τηλεφωνήματα και SMS θέλει να υπάρχουν οροφές και να παραμείνουν οι οροφές αυτές μέχρι το 2016 τα ανώτατα όρια όπως και στους πρώτερους κανονισμούς για την περιαγωγή θέλουμε να μειωθούν τα ανώτατα όρια αυτά. Για εξερχόμενα τηλεφωνήματα περιφέρειων για τον τελικό καταναλωτή, το 2002 θα ήταν 32 ευρώ. Και μέχρι το 2014 θα πρέπει να κατέβει στα 24 ευρώ. Μέγιστη τιμή χοντρική. Λοιπόν, όσον αφορά και τη στοιχεία, όπως αφορά την περιαγωγή, ρυθμίσαμε τη χοντρική τιμή και τώρα θέλουμε στην τελική τιμή να τεθούν ανώτατα όρια και σε αυτόν τον τομέα και τιμές χοντρικής μέχρι το 2014 θα είναι 15 ευρώ ανά 10 και 15 cents ανά megabyte. Και 1η Ιουλίου το 2016 θα κατοργηθούν οι οροφές και ελπίζουμε να έχουν λειτουργήσει μέχρι τότε τα διαθωτικά μέτρα. Λοιπόν, και θα πρέπει να ακολουθήσουμε τη σωστή προσέγγιση θα πρέπει να κινηθούμε και στο επίπεδο των χειριστών του δικτύων που θα πρέπει να μην αρνούνται την πρόσβαση στα δίκτυά τους στους φορείς που δεν έχουν το δικό τους δίκτυο. Ξέρουμε πολύ καλά τα θέματα της, ε, από, του, του unbundling, της αποσυνδέσεως σε άλλους τομείς και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εδώ στο άρθρο 4, Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σαν στόχο την ξεχωριστή παροχή διαδικτύου τηλεφωνίας είναι η αποσύνδεση την οποία γνωρίζουμε και με τη θέση των ανωτάτων ορίων στα τέλη και με τα διαθετικά μέτρα πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει προτάσεις που εντάσσονται στο γενικότερο διάβημα με το οποίο συμφωνώ. Είναι μια καλή προσέγγιση, είναι μια διτή προσέγγιση, οδηγεί σε αύξηση του ανταγωνισμού. Έχω έρθει σε επαφή με τον τομέα, με τους ενδιαφερομένους και όσον αφορά τον τομέα αυτό είναι σημαντικό να μπορούν να βασίζονται στην εμπιστοσύνη των χρηστών Πολύ συχνά υπάρχουν προβλήματα όταν μετακινούνται οι πελάτες στο εξωτερικό, διότι φοβάται ο πελάτης το κόστος της περιαγωγής. Μέσω διευθυντικών μέτρων και των οροφών θέλουμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη, να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη στον τομέα, ούτως ώστε εσωτερική αγορά να πραγματοποιηθεί, να λειτουργεί πραγματικά και να μπορέσουμε να προοδεύσουμε ε, και στον τομέα των διαφόρων προγραμμάτων για την πρόθεση της ψηφιακής τεχνολογίας. Τώρα όσον αφορά τη δική μου αξιολόγηση, θέλω και τη δική σας βέβαια, θα έλεγα ότι όσον αφορά την τηλεφωνία και τα SMS, η πρόταση δεν είναι κακή κατά την απόψή μας. Μπορούμε να ζητήσουμε να δούμε ποια είναι τα περιθώρια ελιγμών. Ίσως μπορούμε να μειώσουμε ακόμα περισσότερο τις οροφές αλλά το σημαντικότερο, αυτό που θεωρώ ότι είναι σημαντικότερο, είναι να έχουμε θέση όσον αφορά την περιαγωγή των στοιχείων. Σε αυτό το τομέα πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ήταν αρκετά φιλόδοξη και θα πρέπει να προχωρήσουμε λίγο περισσότερο, ούτω ώστε να μειωθεί η διαφορά που υπάρχει μεταξύ των αρχικών τιμών και ε, των τιμών τις οποίες καταβάλει ο τελικός καταναλωτής. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το συζητήσουμε. Νομίζω ότι εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε αυτά τα ανώτατα όρια, τις οροφές, όσο τα διαθωτικά μέτρα δεν έχουν λειτουργήσει και δεν είμαστε σίγουροι για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Όσον αφορά τα διαθωτικά μέτρα, θα ήθελα να πω ακόμα το εξής. Πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμόζονται τα διαθωτικά μέτρα Δηλαδή σε ποιο βαθμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθεί ουδέτερη προσέγγιση από πλευράς τεχνολογικής, δείχνοντας κάποιες διεξόδους ταυτόχρονα. Πρέπει να δούμε κατά πόσο η προσέγγιση είναι απλή ή αν υπάρχει κάποια ε, διτή προσέγγιση. Αν χρειαζόμαστε ε, μία δεύτερη κάρτα SIM που να χρησιμοποιείτε στο τηλέφωνο. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μπορέσει να μας πει περισσότερα πράγματα. Αν περνάει κανείς από τον ένα πάροχο υπηρεσιών στον άλλον. Τι γίνεται. Όταν διάβασα αυτό το κείμενο πρώτη φορά θεώρησα ότι δεν αναπόκειται σε μας να ασχοληθούμε με αυτό που αποκαλείται local breakout και τις άλλες τεχνικές στοιχείες που αναφέρονται. Στόχος θα έπρεπε να είναι να έχουμε μια γενική εικόνα όσον αφορά τη δέουσα προσέγγιση για να καταλήξουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το χρήστη. Θα πρέπει να συζητήσουμε και τις λεπτομέρειες. Νομίζω ότι θα έχουμε πραγματικό ανταγωνισμό αν έχουμε τελικά στα χέρια μας ένα μηχανισμό ο οποίος να είναι φιλικός προς το χρήστη. Το σύστημα να είναι φιλικό προς το χρήστη. Ούτως ώστε ο κόσμος να μην λέει πια αν περάσω τα σύνορα θα, με, θα, θα έχω φοβερό λογαριασμό. Εντάξει, συγγνώμη που εκφράζομαι και αναφέρομαι σε αυτά τα θέματα, αλλά πολλοί κόσμοι έτσι αυτό λέει. Θα, θα, πληρώνω, θα πληρώσω πανάκιου λογαριασμού απέναντι στα σύνορα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ρυθμίσει κάτι άλλο. Το θέμα Τον deal bill shocks, δηλαδή το, το ότι έρχεται ο λογαριασμό, ο οποίο ε, είναι τόσο φοβερό που ταράζει τον καταναλωτή πρέπει να πληρώσει. Μήπω θα έπρεπε να προβλέπετε κάποια λύση όσον αφορά και τη μετακίνηση εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πάει κανείς στην Αίγυπτο, στις Ηνωμένες Πολιτείες κλπ. Ε, να του λένε την τάξη μεγέθους δηλαδή να προειδοποιούν τον πελάτη μην, μην πάθει τίποτα. Νομίζω πως είναι μια πρόταση που έγινε από έναν συνάδελφο, δεν ε, την ε, υιοθέτησε η Κομισιόν, αλλά θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους να την υιοθετήσουν. Μετά, με ποιες ε, μονάδες υπολογισμού θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Εδώ πέρα προτείνει κιλομπάιτ, megabyte η Κομισιόν. Ε, μίλησα με τον Κρίστιαν Έγκστρομ των Πρασίνων που λέει πως θα πρέπει πλέον να μιλάμε για gigabyte. Δεν ξέρω εδώ πέρα τι προτιμάτε εσείς. Για εμένα είναι σημαντικό να ακούσω τι άποψη έχετε για τον κανονισμό roaming 3. Εγώ θεωρώ πως είναι καλή η πρόταση της ε, Κομισιόν η οποία μπορεί να βελτιωθεί σε κάποια σημεία. Ο στόχος είναι σαφής ανταγωνισμό να έχουμε στην αγορά και θα πρέπει να έχουμε κατά νου και τη ρύθμιση των τιμών, δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα κίνητρο ε, για να κινητοποιηθούν ε, να μπουν νέες εταιρείε στην ε, αγορά. Βεβαίω θα πρέπει να υπάρχει και μια διαφορά μεταξύ των, των πελατών Λιανικής και των υπολείπων, αλλά να ισχύσουμε και τους πελάτες εδώ πέρα, αλλιώς δεν θα βοηθήσει τίποτα ο κανονισμός. Αυτά για την ουσία. Τέλος για το χρονοδιάγραμμα κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω το συντομότερο δυνατόν να υποβάλω το πρώτο σχέδιο της έκθεσης ε, για να μπορέσουμε ίσως φέτος ήδη σε μία από τις τελευταίες συνεδριάσεις τις φετινές πριν από τα Χριστούγεννα να το συζητήσουμε. Έχω γράψει εδώ πέρα 19 ε, Δεκεμβρίου θα μπορούσαμε ίσως να συζητήσουμε την έκθεσή μου. Καλό θα ήταν να γίνει μία μήνυα ακρόαση Έχοντα κατά νου βεβαίω και την τεχνική εφαρμογή, αλλά όχι μόνο για αυτό το ζήτημα, και μετά να δούμε και την προθεσμία για τις ε, τροπολογίες. Όσο πιο γρήγορα κινηθούμε, τόσο το καλύτερο. Ξέρω πως είναι κάτι το τρομακτικό για όλους μας συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση, αλλά στόχος είναι ο κανονισμός ο τρίτος ε, να συνδεθεί άμεσα με τον κανονισμό τον δεύτερο και θα προσπαθήσω ε, όσο μπορώ για να τα καταφέρουμε για να μπορέσουμε πριν, τις, ε, πριν το καλοκαίρι του επόμενου έτους να στείλουμε το μήνυμα στους καταναλωτές μας πως αυτή η εσωτερική αγορά ε, για το roaming και για όλες τις υπηρεσίες φωνής, SMS και δεδομένων υπάρχει στην Ευρώπη. Αυτά. Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία και σας ευχαριστώ και για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε, Αγγέλικα. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, δύο παρατηρήσεις επί της διαδικασίας. Ε, για τη μήνυα ακρόαση, το είπαμε, θα γίνει γύρω στις 19-20 Δεκεμβρίου και μου λέει η γραμματεία πως... Μετά θα ακολουθήσουν σύντομα οι τροπολογίες, ε, γιατί ούτως ή άλλως θα πρέπει να καταθούν με βάση την πρόταση της Κομισιόν. Οπότε θα προσπαθήσουμε να είμαστε γρήγοροι. Βεβαίως το θέμα είναι το πώς θα το πόσο θα το συζητήσουμε ή όχι. Και βεβαίως η διαφορά εδώ πέρα από τις υπόλοιπες περιπτώσεις είναι πως ε, όσον αφορά την ε, περιαγωγή ε, κατ' ουσίαν συζητάμε τρίτη φορά το ίδιο πράγμα, δεν είναι τίποτα το καινούριο. Θα περιμένω βέβαια να δω πώς θα αντιδράσουν και οι συνάδελφοι. Λοιπόν, η κυρία Ντελκαστίγιο. Ε, ε, Ευχαριστώ. Θα είμαι λακωνική, γιατί είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την αναθεώρηση αναδιατύπωση για το roaming, την περιαγωγή. Είναι πολύ περιεκτική η παρουσίαση που μας έκανε η Αγγέλη Κανίμπλερ της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι ενδιαφέρουσα για να σημειώσουμε κάποια πρόοδο ανάλογα με τις αρμοδιότητές μας για την εσωτερική αγορά. Ακούσαμε από την ανάλυση που έγινε ότι οι τιμές μεν μειώθηκαν, αλλά ανταγωνισμός δεν υπάρχει σε υψηλό επίπεδο. Υπήρξε κάποια συμφωνία σε ό,τι αφορά το ανώτατο όριο μεταξύ των περισσότερων παρόχων υπηρεσιών, αλλά στην ουσία δεν βελτιώθηκε ο ανταγωνισμός. Κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει δεν είναι να επισέλθουμε σε σχολαστική ανάλυση συγκεκριμένων θεμάτων, αλλά να διαμορφώσουμε μια στρατηγική ε, εντύπωση και θέση για την αναδιατύπωση του κανονισμού για το roaming. Κατά τη γνώμη μου, η αναδιατύπωση αυτή, πέραν ε, το, φωνή θα πρέπει, της φωνής να περιοριστεί στα δεδομένα γιατί το, ο δεύτερο κανονισμό roaming, roaming περιοριζόταν στα τηλέφωνα, στη φωνή. Ο τρίτο θα πρέπει να καλύψει τα δεδομένα. Περιαγωγή δεδομένων. Η περιαγωγή, η μεταβίβαση δεδομένων θα πρέπει να γίνεται στα πλαίσια μιας ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς και με υποδομές που θα επιτρέπουν αυτή τη μεταβίβαση. Επίσης, να συνδέσουμε την περιαγωγή με το φάσμα. Ψηφίσαμε τη σχετική έκθεση γιατί έτσι μπορούμε να έχουμε κινητή ευρυζωνία και να βελτιώσουμε την ταχύτητα και τον όγκο μεταβίβασης δεδομένων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το θέμα των υποδομών το έχουμε. Μας λείπει το σκέλος της ανταγωνιστικής αγοράς σε ό,τι αφορά την περιαγωγή και της φωνής, των φωνητικών μηνυμάτων. Και φυσικά να μην ξεχάσουμε και τα δεδομένα, την περιαγωγή δεδομένων. Ο κόσμος ε, εξελίσσεται ραγδαία σε ό,τι αφορά τη μεταβίβαση δεδομένων με ανταγωνιστικούς όρους. Πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να είναι και ο δικός μας στόχος. Η περιαγωγή θα πρέπει την τρίτη αυτή φάση να επικεντρωθεί στη μεταβίβαση των δεδομένων. Αλλά θα πρέπει να σπεύσουμε και να επισέλθουμε κάποια στιγμή και στι λεπτομέρειε των μηχανισμών προκειμένου να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα στην περιαγωγή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκόμες. Γκέμπελ, συγγνώμη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Άντζελικα Νίμπλερ για την πολύ καλή παρουσίαση που μας έκανε ε, και την εισαγωγή στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χάρη στην περιεκτική αυτή παρουσίαση δεν θα χρειαστεί και εγώ να μακρηγορήσω σήμερα. Είχα συνεργαστεί στο παρελθόν με την Αγγέλικα για το πρώτο κανονισμό roaming ε, τότε που ήταν πρόεδρος της Επιτροπής και είχαμε πολύ αποτελεσματικό τριμερή διάλογο και μάλιστα επιβάλαμε, καταφέραμε και ε, επιβάλαμε τις απόψεις του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο. Ήταν σημαντική επιτυχία μας τότε, στον πρώτο κανονισμό ε, της περιαγωγής. Μετά το δεύτερο, και το δεύτερο ρόμιγκ όμως, έχουμε ε, αστρονομικές ε, ακόμη τιμές ε, στην περιαγωγή στην Ευρώπη και όχι μόνο για τη μεταβίβαση των δεδομένων δεν άλλαξε και πολύ σε ό,τι αφορά το ύψος των τιμών. Όλοι όσοι έχουν κινητό και νομίζω ότι όλοι πια έχουμε κινητό, οπότε όλοι στο δύο καζάνι βράζουμε, γνωρίζουμε ότι είναι αδύνατον να διαβάσουμε το, το λογαριασμό του τηλεφώνου. Είναι, είναι ακατανόητα αυτά που περιλαμβάνει ο λογαριασμός δεν είναι καθόλου φιλικός προς το χρήστη. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιωθεί και αυτό το σκέλος για να γίνει πιο ευανάγνωστο ο λογαριασμός. Και φυσικά χρειαζόμαστε την απαραίτητη ενημέρωση για τις τιμές. Μερικοί υπάρχοι υπηρεσιών ε, κάνουν επιθετικές προσφορές για τους νέους πελάτες, αλλά γενικώ έχουν την τάση να ξεχνούν τους παλιούς. Ε, ή δεν υπάρχει κάποια συνέχεια. Θα πρέπει λοιπόν ε, να μεριμνήσουμε ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών να περιλαμβάνουν στις προσφορές τους ε, για τους νέους πελάτες και τους παλιούς και αυτοί να ευνοούνται. Σε ό,τι αφορά την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής πιστεύω ότι βαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση παρόλο που σίγουρα θα χρειαστεί να εξετάσουμε κάποια επιμέρους σημεία. Και σας παραπέμπω εδώ στην ανάλυση του Μπερέκ. Αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες αυτές στη συνάντηση με τους και ηγητές και την Αντζέλικα Νίμπλερ. Πιστεύω ότι θα υπάρξει ευρία συνεργασία μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Το είχα διατυπώσει αυτό και σε μία δημόσια κρόση που είχαμε οργανώσει για το θέμα στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία. Δυστυχώς τα πρώτα θύματα των αστρονομικών απαγορευτικών τιμών που εφαρμόζονται είναι οι ευρωβουλευτές, γιατί οι ευρωβουλευτές είναι οι οι καταναλωτές, οι χρήστες της περιαγωγής και πληρώνουν και την ύφη αυτών των τιμών. Το θέμα είναι αυτό το άνοιγμα προς τον ανταγωνισμό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ευνοήσει όντως και τους νέους ερχόμενους στην αγορά ή τους μικρούς παρόχους υπηρεσιών ή μήπως θα ωφελήσει μόνο τους μεγάλους παρόχους. Εγώ διαπιστώνω ότι η Vodafone, Orange και η Τελεφώνικα και όλες αυτές οι μεγάλες επιχειρήσεις ούτως, ούτως ή άλλως είναι παρούσες σε όλες τις, σχεδόν τις χώρες. Και όταν έρχονται εκπρόσωποι αυτών των μεγάλων ομάδων, ε, μεγάλων επιχειρήσεων, μας λένε ότι τους αρέσει πολύ η ευρωπαϊκή αγορά, αλλά για λόγους ε, τιμών προσπαθούν να ε, προτιμούνται στενά εθνικά σύνορα. Δηλαδή, να κρατήσουμε τη λογική της εσωτερικής αγοράς, αλλά να εφαρμόσουμε μια εσωτερική αγορά γνήσια και για την περιαγωγή και κυρίως για την περιαγωγή δεδομένων. Εκεί είναι που υπάρχουν μεγάλες καταχρήσεις. Απομένει και το ζήτημα των σχέσεων με τις τρίτες χώρες. Όταν ταξιδεύει κανείς στο εξωτερικό και αυτό είναι καθημερινότητα για μας, πολύ συχνά πηγαίνουμε σε αποστολές και μένουμε μερικές φορές ευρώντιτοι όταν παίρνουμε το λογαριασμό. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πώς θα λύσουμε το πρόβλημα. Για να αποφύγουμε και κάποιες ανακοινώσεις ε, που είναι περιττές από τους τοπικούς παρόχους. Αυτές οι ανακοινώσεις ε, πραγματικά δεν μας εξυπηρετούν καθόλου, πολλό δε μάλλον το μερικές φορές χρεώνουν και όλα τις πληροφορίες που μας στέλνουν, χωρίς να τις έχουμε ζητήσει. Ελπίζω να επιταχύνουμε τις διαδικασίες και γιατί όχι να καταλήξουμε και στη συμφωνία με το Συμβούλιο στην πρώτη ανάγνωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βαλεάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα σας ε, παρουσιάσω και εγώ μερικές ε, σκέψεις. Αυτή ε, η αρρύθμιση των κανονισμών το roaming μας δίνει τεράστιες δυνατότητες. Ίσως μέχρι να φτάσουμε στο κανονισμό 15 για την περιαγωγή καταλήξουμε σε προτάσεις που θα είναι αυτές πραγματικά που προσδοκούν από τις υπηρεσίες ε, οι καταναλωτές. Βρισκόμαστε στον τρίτο κανονισμό για το roaming, την περιαγωγή και με την Αντζέλικα είχαμε συνεργαστεί όχι από τον πρώτο κανονισμό της περιαγωγής αλλά και στο δεύτερο ήταν πρόεδρος προέδρευσε σε τριμερείς διαλόγους είχαμε πολύ επιτυχημένους τριμερείς διαλόγους και όλοι είχαμε ελπίσει ότι θα βελτιωθεί η περιαγωγή για τους Ευρωπαίους και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε θα ήθελα να συγχαρώ βέβαια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να πω ότι υποστηρίζω την προσέγγισή της γιατί είναι η πρώτη φορά που προσπαθούμε να θεσπίσουμε κάποια διαρθρωτικά μέτρα. Και ο στόχος εξασφάλισης ανταγωνιστικότητας στην αγορά είναι σημαντικός. Θέλουμε ποιοτικέ υπηρεσίες σε προσιτές τιμές για τους καταναλωτές. Πολύ ωραίοι και αξιέπαινοι στόχοι, αλλά τέτοιους στόχους είχαμε και στο πρώτο κανονισμό και στο δεύτερο κανονισμό για την περιαγωγή. Ήδη από το δεύτερο κανονισμό ζητήσαμε ε, διαρθρωτικά μέτρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τώρα μας τη προτείνει. Πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση, αλλά συνήθω οι, ε, οι προσεγγίσεις είναι διτές, αλλά και οι διπλές αυτές προσεγγίσεις ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση, είναι παράλληλες ε, και έτσι δεν θα δημιουργήσουν σύγχυση. Και το unbundling ιδιοκτησιακός διαχωρισμός χωρίς τη χρέωση. Να δούμε αν αυτή η αποδέσμευση λειτουργήσει. Μακάρι. Οι διαφορές τιμών είναι μεγάλες. Βέβαια, εξακολουθούν να ισχύουν τα ανώτατα όρια και φυσικά τα ανώτατα όρια θα πρέπει να συνοδευτούν από τη μέτρα για την αποδέσμευση σε αυτό το στάδιο. Βέβαια, τα δημαγωγικά μέτρα υπέρ της μείωσης των ανώτατων ορίων, να δεν εφαρμοστούν υπήρξαν κάποια προβλήματα με την περιαγωγή δεδομένων και είδαμε ότι οι τιμές χονδρικής μεν μειώθηκαν, αλλά οι τιμές ελληνική εξακολουθούν να είναι αστρονομικές. Αυτό το ζήτημα θα πρέπει να το συζητήσουμε περαιτέρω. Τα υπόλοιπα είναι ίσονο σημασία, λεπτομέρειες. Θα δούμε αν θα επιλέξουμε απλά, διπλά, IMSI ή ένα συνδυασμό του συστήματος. Πάντως όποια προσέγγιση και διαλέξουμε θα πρέπει να είναι εύχρηστη για τους καταναλωτές. Γιατί αν η λύση είναι περίπλοκη θα καταλήξουμε στο, στη διατήρηση της παρούσας κατάστασης του quo για τους εθνικούς παρόχους. Τώρα αν ταχθούμε υπέρ της αποδέσμευσης ε, της χωρίς της γιατί να μην μπορεί ο καταναλωτής να αγοράσει ε, υπηρεσίες roaming από διαφορετική χώρα από αυτήν ε, στην οποία αγόρασε το κινητό και έχει τις εθνικές υπηρεσίες. Όταν ο καταναλωτής ακούει unbundling, ε, χωρίς τη χρέωση αποδέσμευση, περιμένει μία πανευρωπαϊκή προσέγγιση. Και μια και μιλούμε για το unbundling αυτό, την αποδέσμευση, να δούμε αν θα μπορέσουμε να επιλύσουμε και το πρόβλημα. Αυτά προς το παρόν. Εγώ συνήθως θα υποστηρίξω την πρόταση, θα είμαι συνεργάσιμη και μια και όλο οι ίδιοι ε, μιλούμε για το θέμα αυτό, είμαστε γνωστοί ύποπτοι. Ε, πιστεύω ότι θα βοηθήσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει και νέες φαϊνές ιδέες. Ευχαριστώ. Uh, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Αγγέλικα για την πολύ καλή εισαγωγή. Δεν θα επαναλάβω όσα μας είπες, διότι τίνω να συμφωνώ με τα περισσότερα από αυτά που είπες. Θα έλεγα ότι δεν θέλω να οδηγηθώ σε λαϊκιστικό αγώνα προς τα κάτω όπως η Παντριάννα, αλλά να δούμε αν τα ανώτατα όρια είναι τα ενδεδειγμένα. Και η μεγαλύτερη μου ανησυχία αφορά τα διαθωτικά μέτρα και κυρίως στον τομέα της χοντρικής. Είμαστε σίγουροι ότι αυτό που κάνουμε καλύπτει το θέμα. Αυτό που βλέπω είναι ότι όσον αφορά τη χοντρική, διαισθάνομαι και υπάρχει διαφορά μεταξύ διέστησης και στοιχείων, διαισθάνομαι ότι η προσέγγιση των εμπορευομένων, των εταιριών είναι περισσότερο προσέγγιση καρτέλ. Δηλαδή συμφωνούν μεταξύ τους να μην βλάψουν ένας τον άλλον. Και θα έλεγα ότι αυτά θα έπρεπε να σχετίζονται περισσότερο με να αφορούν τον Επίτροπο, τον υπεύθυνο για τον ανταγωνισμό. Και φοβούμαι ότι χρησιμοποιούμε τα ανώτατα όρια και παρόμοια μέτρα για να αντιμετωπίσουμε αυτό που υποψιαζόμαστε ότι είναι το καρτέλ των μεγάλων εταιριών. Και δεν είναι σωστή προσέγγιση αυτή. Θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε, πιστεύω, την ακρόαση που θα οργανώσουμε για να το ερευνήσουμε σε περισσότερο βάθος. Εάν δεν έχουμε καλύτερη επιλογή από αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ είμαι υπέρ. Αλλά να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα αφήσουμε καμία περίπτωση ανεξερεύνητη. Ίσως να υπάρχουν διορθωτικά μέτρα συμπληρωματικά που θα πρέπει να εξετάσουμε και θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και στο κείμενο. Όχι εις βάρος βέβαια του να καθυστερήσουμε. Άρα και ο χρονισμός είναι πολύ σημαντικός. Θα ήθελα να προτείνω έναν-δύο ομιλητές για την ακρόαση που θέλουμε να διοργανώσουμε, ούτως ώστε να εξεταστεί το θέμα της αγοράς χοντρικής και η ανταγωνιστικότητα ή μάλλον η έλλειψη αυτής. Ο συνάδελφος Τσίτσεστερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ την Αγγέλικα Νίμπλερ για την παρουσίασή της. Έκανε πολλή δουλειά στον τομέα αυτό και είναι καλή δουλειά παρατήρησης. Εμείς όταν θέσαμε τα ανώτατα όρια, δεν πετύχαμε τα αποτελέσματα, δηλαδή την τόνωση του ανταγωνισμού στον τομέα. Και βάσει τον, όπως τον είπε και ο Φίλιπ Λάμπερτς, οι τιμές των εταιριών έτειναν να ανέβουν στην οροφή και να μείνουν εκεί. Άρα δεν καταφέραμε να εισαγάγουμε ανταγωνισμό στον τομέα. Αυτό είναι άκρως απογοητευτικό. Και ο όγκος φωνητικής κυκλοφορίας, για να κάνουμε διαχωρισμό φωνητικής επικοινωνίας και δεδομένων, ε, παρέμεινε στατική, στατικός. Εγώ ήλπιζα όταν ξεκινήσαμε στο δρόμο αυτό, στο Roaming 1, εγώ ελπίζω ότι υποχρώνω τι εταιρείε να μειώσουν τι τιμέ του, ο κόσμο θα ενθαρρυνόταν να χρησιμοποιεί τι δυνατότητε περιαγωγή. Αυτό δεν συνέβη όμω. Ηρίστον παρόδο. Κύριε Γκέμπελς, Α θυμηθούμε ότι αυτό είναι προ όφελο των καταναλωτών, όχι των Ευρωβουλευτών. Διότι ο τομέα μα κατηγορούσε ότι θέλαμε να μειώσουμε τι τιμέ για τη δική μα βολή. Θέλουμε να το κάνουμε αυτό για του εκλογεί μα. Αυτού θέλουμε να βοηθήσουμε περισσότερο από εμά. Συμφωνούμε, συμφωνούμε, λέει και ο Σιτζεστέρ. Να πω λοιπόν ότι μου αρέσει η ιδέα αυτή τη αποσύνδεση, των bundling, δηλαδή και εντός χώρας και εκτός και έτσι πιστεύω ότι θα υπάρξει μεγαλύτερος ανταγωνισμός παρομοίως και διαχωρισμό δεδομένων από, τα, τη φωνητική επικοινωνία. Ελπίζω να μπορέσει η βιομηχανία να ανταποκριθεί σε αυτό και να ανταγωνιστεί μια εταιρεία με την άλλη. Αυτό που είπε η Αγγέλικα τώρα για το, το bill shock, δηλαδή το ότι παθαίνει κανείς σοκ από το λογαριασμό. Κάτι μπορεί να πλήξει τον αθώο καταναλωτή που ταξιδεύει το στο εξωτερικό και του έρχεται μετά ο λογαριασμό και του έρχεται ταμπλά. Ε, μου άρεσε η αρχική νομοθεσία που υποχρέωνε τι εταιρείε να προειδοποιούν τους πελάτες τους όταν έφταναν σε πολύ ακριβό λογαριασμό ή όταν έμπαιναν σε μια κατάσταση περιαγωγής. Και πρέπει να πω ότι νομίζω ότι είναι καλή αρχή που ακολουθήσαμε Δηλαδή να αγοράζεις εν γνώση σου, να σε έχουν προειδοποιήσει. Αυτή είναι η σωστή αρχή που χρησιμοποίησαμε. Διότι θα πρέπει οι άνθρωποι να, έχουν την, να αναλάβουν την ευθύνη για τις αποφάσεις του τι αγοράζουν και τι δεν αγοράζουν. Λατινιστή, caveat emptor. Λοιπόν, πρέπει να προστατεύσουμε τους καταναλωτές από αυτό το, από αυτή την πιθανότητα. Πώς? Να δημιουργήσουμε ένα δικαίωμα έφεσης για τους καταναλωτές να μπορούν να προσφύγουν στην Εθνικό, Εθνική Ρυθμιστική Αρχή σε κάποιον, αν θεωρήσουν ότι ο λογαριασμό του είναι υπερβολικό. Δύσκολο να καθοριστεί αυτό, το δέχομαι. Τι είναι υπερβολικά, τι αποτελεί υπερβολικά μεγάλο λογαριασμό, Αν κάποιο την έχει πατήσει όμω, ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. το θέτω σαν δυνατότητα αυτή, σαν πιθανότητα. Διότι θα κάνω ακόμη πιο ριζοσπαστική πρόταση. Σε λίγο θα την ακούσετε για τη φωνητική περιαγωγή. Ίσως βρούμε έναν τρόπο για να επιφέρουμε πειθαρχία επί των εταιριών. Εκτός πέρα από το να θέσουμε το νοτοτόριο σε εναλλακτική λύση. Η ριζοσπαστική μου λύση. Λοιπόν, για την ε, φωνητική περιαγωγή προσέγγιση μας δεν λειτουργήσε. Έχω επιφυλάξει σοβαρές όσον αφορά την παρέμβαση στην αγορά. Και επι, επιβάλλοντας τιμές αυτό είναι κάτι που δεν είναι ανταγωνιστικό. Εάν υπάρχει κατάξυση αγορά, δικαιολογείται. Όπω γινόταν παλιά με τι εταιρείε όσον αφορά την περιαγωγή και τα τέλη που επέβαλαν. Μπορούμε να επανεξετάσουμε το θέμα. Μήπω ήρθε η ώρα να δώσουμε στι εταιρείε μια δεύτερη ευκαιρία. Πώ. Αφαιρώντας τι ανώτατες τιμέ, τα ανώτατα ωρία όσον αφορά τη φωνητική περιαγωγή και ταυτόχρονα, όπως είχαμε εισαγάγει και την αποσύνδεση, τον bundling, να πούμε είπατε ότι μπορείτε να ανταγωνιστείτε. Επανειλημμένα μας είπαν αυτό το θέμα. Μπορούμε να ανταγωνιστούμε, μην μας δίνετε όρια. ωραία, λαμπρά. Κοιτάξτε, ας το σκεφτούμε το εξή. Να τους δώσουμε μια περίοδο χάριτος, ας πούμε. Δεν έχετε ανώτατα όρια. Αλλά αν το καταχραστείτε αυτό και δεν ανταγωνιστείτε, θα ξαναφέρουμε τα ανώτατα όρια. Ε, το ρίχνω στο τραπέζι αυτό σαν πρόταση εναλλακτική προσέγγιση. Διότι εγώ βλέπω ότι δεν πετύχαμε. Και προσπαθούμε να ελέγχουμε όλο και περισσότερο τις τιμές και να είμαστε όλο και πιο παρεμβατικοί. Και αυτό αντιβαίνει τους στόχους, τους επιδιωκόμενους της ενιαίας αγοράς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Thanks, Ευχαριστώ Ρούμπιχ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την Αγγέλικα Νίμπλερ. Δεν πιστεύαμε όλοι πως χρειαζόμασταν και τρίτο κανονισμό για το roaming. Θα έπρεπε να έχει λυθεί με τον πρώτο κανονισμό το πρόβλημα, αλλά αυτό πιστεύω μας δείχνει την πραγματικότητα. Πως η τεχνική πρόοδος δηλαδή είναι πάρα πολύ δυναμική και είναι αναγκαίο να προσαρμόσουμε τις συνθήκες πιο σύντομα. Και χρειάζεται αυτό για αυτές τις δραστηριότητες. Για εμάς πολιτικούς δεν είναι σημαντικό μόνο να μπορούμε να αποδείξουμε στους πολίτες μας πως είναι πράγματι δυνατό να δημιουργήσουμε μια κοινή αγορά. Πάρα πολλές ε, εταιρείε το θέλουν επίσης και θέλουμε να αποδείξουμε πως είναι δυνατό μέχρι το 2014 γιατί βεβαίως ε, τότε θα κριθούμε ως πολιτικοί σε επόμενες ευρωεκλογέ και θέλουμε και από την Κομισιόν μια έκθεση μέχρι τότε για το πώς λειτουργεί και τι έχει επιτύχει ο κανονισμός αυτός για τους πολίτες της Ευρώπης. Νομίζω πως αυτό είναι το αποφασιστικό. Είδαμε πως είναι ένα θέμα το οποίο είναι γνωστό στους πολίτες της Ευρώπης. Πρέπει επίσης να συζητήσουμε πώς θα ενισχύσουμε την ε, διαφάνεια και για την, ε, θα πρέπει να μπορούν να βλέπουν και τη, το ποσό και την τιμή ανά μονάδα βεβαίως θα πρέπει λοιπόν να δοθούν εδώ πέρα επιπρόσθετες πληροφορίε ε, ποια είναι η ποσότητα των δεδομένων, ποιο πόσα λεπτά έχει χρησιμοποιήσει κανεί ποια είναι η τιμή για όλα αυτά, πόσο τη εκατό του πακέτου του. Νομίζω πω ε, είναι πολύ καλή η θέση εδώ πέρα των εταιριών περί διαφάνειας. Επίσης, θα πρέπει η μονάδα υπολογισμού να παραμένει το kilobyte ε, πράγματι, αλλά οι τιμές ε, θα μπορούσαν να οριστούν ε, σε gigabyte, στη λιανική και βέβαια στη χοντρική σε terabyte. Γιατί τα δίκτυα LTE και τέταρτης γενεάς ε, θα οδηγήσουν σε τελείως διαφορετικές ποσότητες δεδομένων. Δηλαδή θα μπορεί κανείς να δει ταινίε. Οπότε φαντάζεστε πώς θα λειτουργεί αυτό. Οπότε θα πρέπει να δημιουργηθεί μια δυνατότητα και να στηρίξουμε την Κομισιόν, να δούμε πώς θα μπορέσουμε στην χοντρική αγορά των τηλεπικοινωνιών να περάσουμε στο βήμα, να εγγυηθούμε τη σύνδεση LTE και Wi-Fi. Νομίζω πως είναι σημαντικό να μπορούν να λάβουν μόνες τους οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών ε, την απόφαση πότε μια συσκευή είναι στο Wi-Fi και πότε είναι στο LTE και στο δίκτυο τρίτης γενιάς. Αυτά είναι σημαντικά και βεβαίως ε, όταν ε, μιλάμε για τα SMS να υπάρχει και επιβεβαίωση παράδοσης. Και δεν νομίζω πως χρειάζεται εδώ πέρα μια ε, προειδοποίηση για το SMS. Όσον αφορά τη Λιανική, σημαντικό είναι, βλέπετε εδώ πέρα πως υπάρχουν πάνω από 80 εταιρείε στην Ευρώπη και θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερη επιλογή και μέσω του διαδικτύου και όχι όπως παραδείγματο χάρη στην ε, Ιταλία όπου πρέπει να έχει κανείς ε, ένα νούμερο από το Υπουργείο Οικονομικών και είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά να έχει πρόσβαση στην αγορά. Επίσης, να μην έχουμε αυτές τις λεγόμενες πρόσφορες των συσκευών, αλλά αντιθέτως όπως πάλι και στην Ιταλία να αναφέρονται αναλυτικά όλες οι χρεώσεις, και το κόστος συμβολίων κτλ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ουλσκοκ. Ε, <clears throat> Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πρόταση από πολλές απόψεις είναι θετική γιατί προσπαθεί να αντιμετωπίσει την παράλογη κατάσταση που επικρατεί στην αγορά περιαγωγής και πολύ χρήσιμη ήταν και η εισαγωγή που μας έκανε η κυρία Νίμπλερ. Σε ό,τι αφορά τα διαρθρωτικά μέτρα, ισχύει το ίδιο και εκεί. Χαιρόμαστε για την αύξησή τους, αλλά να μην ξεχνούμε και τις ε, επιφυλάξεις των Ευρωβουλευτών για το ποιες είναι οι πραγματικές πιθανότητες ε, για αυθεντικό ανταγωνισμό στην αγορά. Αυτό μας ενδιαφέρει, ο γνήσιος ανταγωνισμός. Αλλιώς ε, προστεί τα διαφορετικά μέτρα. Σε ό,τι αφορά τα ανώτατα όρια τιμών, φυσικά αυτά τα ε, ανώτατα όρια θα πρέπει να είναι όσο πιο χαμηλά γίνεται. Και να ισχύουν και για τους χρήστες ε, smartphone. Θέλουμε κανόνες που θα προσαρμόζονται και στο σερφάρισμα με κινητό γιατί στο μέλλον θα είναι πολύ πιο γενικευμένο αυτό το φαινόμενο και θα πρέπει περισσότερο προσανατολισμένοι προς το μέλλον να είμαστε και όχι στην κατάσταση των τελευταίων ετών. Γιατί αν χρειαστεί να κάνουμε αξιολόγηση σε ό,τι αφορά την κατάρτιση προτάσεων για τιμές για τις ανώτατες τιμές, ανώτατα όρια τιμών. Πολλές φορές αυτά τα ανώτατα όρια είναι πολύ ψηλά για ένα γιγαμπάιτ θα χρειαστεί να πληρώσουμε 900 ευρώ το 2012 και 700 το 2013 και 500 μετά το 2014 μέχρι το 2016. Αλλά και αυτές οι τιμές είναι υπερβολικές σε μια κοινωνία που εξελίσσεται ραγδαία και σε μια τεχνολογία που εξελίσσεται ραγδαία. Συμφωνώ με τον κύριο Γκέμπελ που είπε ότι καλό θα είναι η προσέγγιση μα να είναι ευρύτερη και να λάβει υπόψη και το καταναλωτή. Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο οι τιμέ, αλλά και η μεταχείριση του πελάτη, ο τρόπο που λαμβάνει τι πληροφορίε. Και φυσικά ευανάγνωστα τιμολόγια, ευανάγνωστοι λογαριασμοί ενδιαφέρον τον καταναλωτή. Γιατί μερικέ φορέ είναι τελείω αποκρυφιστικοί και δυσνόητοι αυτοί οι λογαριασμοί. Κάτι άλλο που μας που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε ποια λογική ισχύει για το επιχείρημα της θέσπισης ανώτατων τιμών των αναφλίων. Γιατί φαίνεται ότι αντί να προσανατολισόμαστε στο μέλλον, κοιτάμε προς το παρελθόν. Ο κύριος Χέκμαρκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι λογικό να αισθανόμαστε εκνευρισμένη και απαγοητευμένη για την κατάσταση στην αγορά αυτή τη στιγμή. Κύριε Ρόιλε, ε, μάλλον βλέπω τον αντιπρόεδρο που είναι Δανός. Όταν τον επισκέφτομαι στη Δανία, στην Κοπεχάγη, και τηλεφωνήσω στη Σουηδία από τη Δανία, από την Κοπεχάγη, θα πληρώσω τα μαλλιά της κεφαλής μου και το σέρφινγκ μέσω διαδικτύου. Αν έρθει όμως ο συνάδελφος ο Δανός στο Μάλμε και τηλεφωνήσει στο Λούλαντ που είναι 800 χιλιόμετρα βόρειος, ισχύει ένα καταποκοπή ποσό. Εκεί δεν θα πληρώσω τίποτα. Παράδοξο αυτό, παράδοξη κατάσταση και πολύ εκνευριστική και απογοητευτική. Δείχνει τις αδυναμίες που, ε, που υπάρχουν στην αγορά. Η αγορά της περιεγωγής και των κινητών είναι η πιο σύγχρονη ε, αγορά του κόσμου και αντί να έχουμε μία μία αγορά, έχουμε 27 διαφορετικές αγορές. Και ακούτε επιχειρήματα, αλλά ε, εδώ έχω την αίσθηση ότι ε, είμαστε ακόμη στην εποχή των, της ασπρόμαυρης τηλεόρασης. Είναι απειρχιωμένο το σύστημα των εθνικών τρόπων συστημάτων περιαγωγής. Είναι σαν την ασπρόμαυρη τηλεόραση. Τελείως παλαιομοδίτικο και παροχημένο. Και είναι πρόκληση και για τους παρόχους υπηρεσιών, και για μας. Θα πρέπει επιτέλους να απαλλαγούμε από το κυρίως πρόβλημα. Αλλιώς θα ε, συζητούμε ατέρμονα για ανώτατα όρια τιμών. Και αλλαγέ ε, δεν θα υπάρχουν αισθητέ. Θα πρέπει να τροποποιηθεί το σύστημα, να έχουμε ενιαία αγορά σε αυτό. Είχαμε ανέκαθεν πρόβλημα με τα ανώτατα όρια τιμών και ο κύριος Λάμπερτ το επισήμανε και ανέφερε και το όρο του ολιγοπολίου καρτέλ. Ε, τα ανώτατα όρια τιμών είναι που δημιουργούν τα ολιγοπόλια, τα καρτέλ, γιατί νομιμοποιούν μία πάγια τιμή. Και αυτό είδαμε, ότι οι τιμές τελικά δεν μειώθηκαν παρά τα ανώτατα όρια. Ευχαριστώ την Αντζέλικα για την παρουσίαση που μας έκανε, γιατί εγώ είμαι υπέρ μιας νέας και πιο σύγχρονης προσέγγιση Ευρωπαϊκή Επιτροπής, που θα λαμβάνει υπόψη και το unbundling, την αποδέσμευση και πολλά άλλα θέματα. Πάντω το έργο αυτό και η Αντζέλικα έχει γνώση και αρμοδιότητα γιατί ασχολείται με τι τηλεπικοινωνίες. Όταν μιλούμε για τον ανταγωνισμό δεν έχουμε μόνο υπόψη τι τιμέ, αλλά και την τεχνολογία. Αναφέρθηκε και το ασύρματο. Ε, αν το σκεφτούμε καλά, μπορούμε εδώ στο Κοινοβούλιο να κάνουμε τηλέφωνα υπεραστικά και υπάρχουν διάφορες εφαρμογές αλλά μερικές φορές ε, το πρόβλημα το παρακάμπτουμε. Θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι ε, στη νέα νομοθεσία δεν επαναλαμβάνουμε τα παλιά προβλήματα, αλλά μένουμε ανοιχτοί προς ε, νέες λύσεις και επιχειρηματικά μοντέλα και αξιοποιούμε και τις ευκαιρίες, τις νέες ευκαιρίες. Και χαίρομαι για την ε, θετική υποδοχή που είχε η νέα πολιτική για το φάσμα συχνοτήτων. Τώρα ανοίγουμε το φάσμα συχνοτήτων και ε, ανοίγουμε και νέες ευκαιρίες, και για πανευρωπαϊκές άδειε. Να αντιμετωπίσουμε το δανέο ειδικό πρόβλημα και άλλα προβλήματα ή να έχουμε άνοιγμα προς νέες τεχνολογίες. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Γι' αυτό, στην περίπτωση αυτή και στον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε αυτό το κανονισμό θα πρέπει να αναχαιτίζουμε άλλες εξελίξεις αλλού. Θα πρέπει να θετήσουμε μία ανοιχτή προοπτική και να σκεφτούμε ότι η κατάσταση που έχει τώρα είναι σαν την ασπρόμαυρη τηλεόραση, τόσο παροχημένη. Και θα πρέπει από την ασπρόμαυρη να περάσουμε στην έγχρωμη τηλεόραση το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστώ. Ε, eh, eh, ναι, κύριε Πρόεδρε, τώρα αν ζούμε στο παρελθόν, το σήμερα ή το αύριο και τα περί ασπρόμαυρης τηλεόρασης. Πράγματι και εγώ θεωρώ πως ε, συζητάμε για ένα σύστημα στο οποίο μας έχουν ε, εξαναγκάσει. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει να μιλάμε ε, ανώτατες τιμές. Εάν θέλουμε μια πραγματική εσωτερική αγορά στην Ευρώπη, θα πρέπει να έχουμε μια αγορά όπου δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ εθνικής και ευρωπαϊκής κλήσεις και χρέωσης. Υπάρχει μία ενιαία ευρωπαϊκή αγορά με ευρωπαϊκές τιμές. Και να μην έχει διαφορά αν μιλάει κανείς στην Ολλανδία, Βέλγιο ή στο Στρασβούργο. Παντού πρέπει να πληρώνω το ίδιο. Οπότε, όταν το κοιτάω αυτό, αναρωτιέμαι και για τα πλαφόν τα οποία καταργούνται στη Λιανική του 2013 δεν υπάρχει αξιολόγηση του πώς λειτουργήσαν στην, ε, το τι επίδρασκαν στην αγορά. Μήπως θα έπρεπε να το αξιολογήσουμε αυτό. Ίσως θα έπρεπε λοιπόν να συνεχίσουμε με αυτό το σύστημα και δεν υπάρχει επίσης καμία εγγύηση για το ότι θα είναι μετά χαμηλότερη η τιμή και αν υπάρχει προστασία για τον καταναλωτή. Επίσης να ρωτήσω και εγώ καταναλώτρια είμαι επίσης ε, και βρίσκομαι σε αυτή την θέση με το συνεχές ε, roaming. Κοιτάξτε, πρέπει να δει τα διάφορα συμβόλαια ο καταναλωτής ε, και τι γίνεται. Κάποιο είναι φτηνότερο για κάποιες χώρες, κάποιο για κάποιες άλλες, αλλού οι Ηνωμένε Πολιτείε, αλλού η Ασία. Υπάρχει δηλαδή διαφάνεια για να κάνει πραγματικά τις επιλογές του ο καταναλωτής. Κατόπιν. Συμφωνώ και με τον κύριο Λάμπερτ ε, για το να έχουμε ε, για το ότι θα έχουμε τελικά ένα σύστημα καρτέλ εδώ πέρα από την άλλη πλευρά ενώ θα πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός και ανοιχτή αγορά. Και η διαφορά μεταξύ λιανικής και χοντρικής είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εγώ δεν λέω να πούμε ποιες θα είναι τιμές, αλλά είναι τεράστιο το περιθώριο εδώ πέρα. Και μήπως θα πρέπει να υπάρχει ένα επίπεδο προστασίας επίσης για τους ανήλικους. Γιατί είναι αυτοί οι οποίοι καθόλου δεν ασχολούνται με την διαφάνεια των τιμών και είναι οι μεγάλοι χρήστες όλων των ψηφιακών αυτών υπηρεσιών και καταλήγουν οι λογαριασμοί στους γονείς τους. Ευχαριστώ. Η κυρία Τικάου. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κατά την άποψή μου, το ότι προσεγγίζουμε εκ νέου ένα κανονισμό για την περιαγωγή ε, είναι κάτι σημαντικό. Πρέπει να βελτιωθεί ο ανταγωνισμός της αγοράς. Εφόσον δεν έχουμε ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά όσον αφορά τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, είναι κάτι αναγκαίο. Αλλά ίσως η προσπάθεια να είναι επίπονη. Ε, δυστυχώς οι τιμές διαφέρουν από χώρα σε χώρα στην Ευρώπη για να έχουμε κοινή εσωτερική αγορά χρειάζεται σύγκληση ε, τιμών όσον αφορά την κινητή τηλεφωνία. Σύγκληση και των εθνικών τελών αλλά και των τιμών της περιαγωγής και θα πρέπει αυτό να καλύπτεται από τον κανονισμό μας. Συμφωνώ με την αναθεώρηση του κανονισμού όμως πρέπει να, να αποφύγουμε ήδη τώρα εκ των προτέρων να καθορίσουμε ε, τα ανώτατα όρια των τιμών ή τουλάχιστον ένα επίπεδο πέρα από το οποίο αρχίζει να καταργείται αυτό το όριο. Χρειάζεται μια ρήτρα αναθεώρησης ε, πριν ληφθεί κάποια συγκεκριμένη απόφαση για την κατάργηση αυτού του μέτρου. Και η ποιότητα των υπηρεσιών παίζει μεγάλο ρόλο. Πρέπει να εξασφαλίσουμε το ότι ο κανονισμός θα επιτρέψει την ανάπτυξη και διατήρηση και συντήρηση των καταλήλων υποδομών. Να επιτρέπεται η είσοδος στην αγορά νέων εταιριών, αλλά και οι φυστάμενες υποδομές να αναπτυχθούν και να συντηρούνται. Άρα χρειάζονται επενδύσεις και εκείνοι που είναι ιδιοκτήτες των υποδομών θα πρέπει να καταβάλουν σχετικώς προσπάθειες και θα πρέπει να υποστηριχτούν να υποστηριχθεί η συντήρηση των υποδομών. Και τα κριτήρια επιδόσεων με βρίσκει σύμφωνη, το τόνισε και το υπογράμισε ο κ. Ρούμπικ. Δεν θα ήταν αποδεκτό να έρχεται ένα SMS πολλές μέρες αργότερα μετά την αποστολή του Χρειάζονται λοιπόν κριτήρια επίδοσης όσον αφορά την παραλαβή από τον παραλήπτη ενός μηνύματος που έχει αποσταλεί, ενός SMS που έχει αποσταλεί. Χρειάζονται σαφέστατες διατάξεις όσον αφορά το ρόλο των ρυθμιστικών αρχών διότι θα πρέπει οι παρεμβολές να εξαλειφθούν και θα πρέπει οι σχετικές αρχές να παρεύουν. Υπάρχουν αυτές οι παρεμβολές, υποφέρουν οι χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ συχνά κοντά στα σύνορα. και στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και οι χώρε Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν έχουν συγκεκριμένα μέτρα όσον αφορά τα νοτατόρια των τιμών. Χαιρετίζω την προσέγγιση της κυρίας Νίμπλερ. Πιστεύω ότι όλοι θέλουμε να έχουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό τομέα όσον αφορά τι υπηρεσίε. Είναι μελλοντικό τομέα και όλο και περισσότερε νέε υπηρεσίε θα παρέχονται. Υπάρχει και όλο και μεγαλύτερη ζήτηση από πλευρά των χρηστών έχουμε νέα αιτήματα, νέες απαιτήσει και θα πρέπει να προτείνουμε στους καταναλωτές ε, τα σωστά μέτρα, τα σωστά προϊόντα, να τους δίνουν τις σωστές πληροφορίες και θα πρέπει οι εταιρείε να εξελίσσονται σε αυτή την αγορά, η οποία αγορά θα πρέπει να ορθή. Θα πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός και θα πρέπει να υπάρχουν εγγύσει για τι σωστέ συνθήκε για τη διατήρηση και σωστή λειτουργία των ε, δικτύων να δώσω το λόγο στην Κομισιόν εάν ε, συμφωνείτε. Και Τερέρα έχετε το λόγο. Και ε, να πείτε κάτι πριν έρθει η κυρία Επιτροπός. Thank you, thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα σχόλια. Χαίρομαι που ακούω πως υπάρχει στήριξη για τη νέα αυτή προσέγγιση για τα διαρθρωτικά αυτά μέτρα. Πράγματι, ο κανονισμός περιπλαφών δεν έλυσε τα προβλήματα ανταγωνισμού στην αγορά roaming και πρέπει να σκεφτούμε εναλλακτικέ. Και θεωρούμε πως η λύση αυτή είναι μια εναλλακτική. Βεβαίως τώρα υπάρχει μια συζήτηση για το ποια θα είναι η σωστή τεχνική λύση και μήπως θα έπρεπε να την ορίσουμε με λεπτομερία στον κανονισμό. Στην πρότασή μας δίνουμε ένα παράδειγμα γιατί θεωρούμε πως η διπλή αυτή τεχνική λύση θα δώσει μια ευκαιρία για να μπουν νέε εταιρείε στην ε, αγορά της περιαγωγής αλλά και οι υπάρξεις εταιρείες να μπουν σε άλλες χώρες ε, ως πάροχοι μόνο περιαγωγής. Αλλά βεβαίως ε, αυτό δεν αποκλείει άλλες εναλλακτικές. Απλά σημαντικό είναι οποιαδήποτε λύση υιοθετήσουμε τελικά ε, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να επιτρέπει την εύκολη είσοδο στην αγορά και ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι όσο δυνατόν πιο εύκολη για να υιοθετηθεί από τους τελικούς χρήστες. Αυτά τα κριτήρια είναι σημαντικά και πρέπει να επιτρέπει είσοδο, όπως είπα στην αγορά, και ταυτόχρονα να δίνει τη δυνατότητα ανταγωνισμού με τις υπάρχουσες εταιρείε και να δίνει στους καταναλωτές ε, εύκολη πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες από εναλλακτικούς παρόχους. Υπάρχουν ε, και άλλες λύσεις. Είμαι σίγουρος πως έχετε ακούσει τις ε, περισσότερο. Ε, πέρα από το διπλό ύμψη υπάρχει και η λύση του λεγόμενου μονού ύμψη και άλλες λύσεις που αυτή τη στιγμή συζητάμε. Νομίζω η κυρία Βαλεάν ρώτησε αν είναι δυνατόν να επιλέξει κανείς ποιος, ποια εταιρεία θα κάνει περιαγωγή σε μια άλλη χώρα. Υπάρχουν λύσεις νομίζω που μπορούν να εφαρμοστούν, ειδικά για τα δεδομένα. Κυρία Νίμπλερ ρώτησε τι θα σημαίνει η εφαρμογή του unbundling, αν θα πρέπει να αλλάξουμε κάρτα SIM, τι σημαίνει στην πράξη. Με την ε, λύση διπλίου ίμψη πράγματι πρέπει να αλλάξει κάρτα SIM Πρέπει να υπάρχει δηλαδή μια κάρτα SIM με αυτή την δυνατότητα. Οπότε θα πρέπει να αλλάξει η κάρτα στην αρχική φάση υιοθέτηση ε, της λύσης αυτής. Όσον αφορά άλλες λύσεις όπως το ενίο ίμψη, εκεί πέρα δεν υπάρχει ανάγκη τέτοια για να αλλάξει η κάρτα SIM. Υπάρχει ένα ίμψη που θα χρησιμοποιεί και το δίκτυο στο οποίο ανήκει ο καταναλωτής και το εναλλακτικό δίκτυο περιαγωγής. Όταν εξετάζουμε αυτές τις διαφορετικές λύσεις, το θέμα είναι ποια λύση δίνει δυνατότητες ανταγωνισμού σε εναλλακτικούς παράγους και εδώ πέρα βεβαίω υπάρχουν οι διαφορές που θα πρέπει οπωσδήποτε να συζητήσουμε αργότερα. Μετά, για τις για τα πλαφόν στις τιμές και αν είναι σωστό επίπεδο. Πρέπει την πρόταση αυτή να τη δούμε ως ένα πακέτο μέτρων. Έχουμε τα διαρθρωτικά μέτρα, στόχος των οποίων είναι η εισαγωγή του ανταγωνισμού και βέβαια ταυτόχρονα πρέπει να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα των καταναλωτών θέλουμε να δώσουμε κίνητρα σε νέε εταιρείε να μπουν στην αγορά, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν θέτουμε το πλαφόν. Εάν είναι πολύ χαμηλό το πλαφόν, τότε προφανώς δεν υπάρχει κίνητρο οι αναλλακτικέ εταιρείε να μπουν στην αγορά και αυτή είναι η αφετηρία μας. Προφανώς Υπάρχει αρκετός ενθουσιασμός για να κατέβουν, να μειωθούν ε, τα διάφορα πλαφών κατανάλωσης δεδομένων. Και βεβαίως θα αντιμετωπίζει ο κόσμος σοκ ε, με το λογαριασμό, ακόμα και αν έχουμε καταργήσει το όριο, αλλά πρέπει να έχουμε κατά νου πως ε, η αγορά αυτή είναι η πιο δυναμική αγορά roaming. Δηλαδή σε σύγκριση με τη φωνή και τα SMS τα δεδομένα είναι τα πιο δυναμικά και θα πρέπει να προσέξουμε να μην ε, διαταράξουμε τις εξελίξεις ε, και στην αγορά της περιαγωγής και στην ε, εγχώρια αγορά δεδομένων σύντομα κατόπιν για πιθανό καρτέλ η συνεργασία μεταξύ εταιριών ε, στον καθορισμό των τιμών. Νομίζω πως ο κύριος Χέκμαρκ είπε το σωστό. Το πλαφόν στην τιμή είναι κάτι που διευκολύνει τον συντονισμό ε, μεταξύ των εταιριών. Οπότε ξέρουν ποιο είναι το maximum και είναι εύκολο να ευθυγραμμιστούν σε αυτό ακριβώς <coughs> το επίπεδο ή λίγο χαμηλότερα. Και άρα νομίζω πως είναι σημαντικό να επενδύσουμε στο δομημένο σύστημα για να φύγουμε από τα πλαφόν γιατί μετά δεν θα δώσουμε στις εταιρείε αυτό το σημείο να εστιάσουν και να ορίσουν εκεί ακριβώς τις τιμές. Τώρα για το αίτημα περισσότερης διαφάνειας και την δυνατότητα επέκτασης του μέτρου για να καλύπτει και τις υπηρεσίες εκτός Ευρώπης όπως προτάθηκε είναι μια καλή ιδέα κάτι πρέπει να δούμε πιο λεπτομερώς ως ιδέα νομίζω όλοι μπορούν να το στηρίξουν πρέπει να δούμε πως ε, ταιριάζει με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού γιατί είναι αυτή τη στιγμή ένα γενικό μέσο της αγοράς και άρα ισχύει μόνο για το εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ε, ξέρω πώς μπορούμε νομικά να το επεκτείνουμε και για περιαγωγή εκτός της Ένωσης. Και εδώ πέρα θα ολοκληρώσω. Σας ευχαριστώ και πάλι για τα σχόλια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δίνω το λόγο πάλι στην Αγγέλικα Νίμπλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτώντας και την ώρα θα είμαι σύντομη. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις ιδέες, παρατηρήσεις που ακούστηκαν αλλά και για τις πρώτες αξιολογήσεις για την πρόταση της Κομισιόν. Νομίζω σε κάποιους τομείς έχουμε μια βασική συμφωνία, ότι θέλουμε περισσότερο ανταγωνισμό, ότι θα πρέπει να κρίνουμε την ε, πρόταση από τη σκοπιά του καταναλωτή. Τώρα δεν θα μπω στις λεπτομέρειες κύριε Πρόεδρε, αναφέρθηκαν. Νομίζω πως ε, στις περαιτέρω διαπραγματεύσεις με τους κοιόδης ηγητές ε, θα τα ξεκαθαρίσουμε. Ακούω πως η 20 Δεκεμβρίου είναι μια καλή ημερομηνία για τη μήνυα ακρόαση για να έχουν και οι καταναλωτές μια απλή πρόσβαση σε εναλλακτικού παρόχους. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα γίνει και η τεχνική ε, εφαρμογή. Σας ευχαριστώ λοιπόν, σημείωσα πάρα πολλά πράγματα, θα τα λάβω υπόψη και αναμένω την περαιτέρω συζήτηση με τους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ όλοι όσοι συμμετείχαν. Τώρα για την προθεσμία δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Θα προσπαθήσουμε να γίνει ακρόαση το Δεκέμβριο. Οπότε θα πρέπει οι ομάδες να στείλουν τις προτάσεις τους για να έχουμε λίγους αλλά καλύτερους εμπειρογνώμονες. κυρία Νίμπλερ είπε πως θέλει να υποβάλει το σχέδιο έκθεσης τον Δεκέμβριο θα δούμε πότε θα έχουμε την προθεσμία για τι τροπολογίες. Τελειώνουμε με αυτό το θέμα τη ημερήσιας διάταξη και μετά περνάμε με το επόμενο θέμα. Ακούσουμε την κυρία Χέντεγκαρ, την κυρία Επίτροπο, η οποία μπαίνει στην αίθουσα και θα συνεχιστεί η συζήτηση. Machst Betreuung von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 So, liebe Αγαπητοί συνάδελφοι, καλωσορίζω στην Επιτροπή μας για πολλωστή φορά την κυρία Χέντεγκαρντ, αρμόδια για την πολιτική του κλίματος. Ήδη αρκετές φορές είχαμε την ευχαρίστηση να συζητήσουμε μαζί της και έχουμε κάποια γεγονότα τις επόμενες εβδομάδες και μήνες που καθιστούν αναγκαίο να ξανασυνομιλήσουμε μαζί της για να δούμε πώς θα δράσουμε από κοινού και αυτό είναι βεβαίω ενδιαφέρον της Επιτροπής μας. Οπότε σας ευχαριστούμε για το ότι ήρθατε και για το ότι θα μας παρουσιάσετε τις ε, σκέψεις σας. Καλώς ήρθατε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη. Είναι μεγάλη χαρά για μένα που εμφανίζομαι πρώτη επιτροπή σα για μια ανταλλαγή απόψεων Γνωρίζω ότι σήμερα βασικά ενδιαφέρεστε να ακούσετε περισσότερα για τις προοπτικές όσον αφορά τη διάσκεψη για το κλίμα του Ντέρμπαν, αλλά θα ξεκινήσω με κάποιες παρατηρήσεις στο πλαίσιο του διαθρωμένου διαλόγου όσον αφορά το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εθετήσει το πρόγραμμα εργασιών για το 2012 την επόμενη Τρίτη και ο πρόεδρος Μπαρόζο θα παρουσιάσει το πρόγραμμα αμέσως αφού εγκριθεί στην Ολομέλεια. Η καταπολέμηση τη αλλαγή του κλίματο παραμένει μία από τι προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για το 2012. Αυτό το τόνισε και ο Πρόεδρος Μπαρόσο στην πρόσφατη ομιλία του όσον αφορά ε, την κατάσταση κατή στην Ένωση. Είπε και παραθέτω ότι βιώσιμε θέσει απασχόληση θα έρθουν να εστιαστούμε στην καινοτομία και νέε τεχνολογίε συμπεριλαμβανομένων των πρασίνων τεχνολογιών. Πρέπει να δούμε ότι το πράσινο και ανάπτυξη ε, πάνε μαζί είναι μια διτή πρόκληση που αντιμετωπίζουμε και πράγματι είμαι πεπισμένη κατά πολέμηση των αλλαγών του κλίματο και οικονομική ανάπτυξη υποστηρίζουν το ένα το άλλο. Ο πρόεδρο επίση ήταν σαφή στην επιστολή του προ τον πρόεδρο Μπούζεκ μαζί με την ομιλία που έκανε για την κατάσταση στην Ένωση ότι το μελλοντικό ο μεθοδικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι το κλειδί για να πετύχουμε τους στόχους μας στο κλίμα. Μπορούμε να κάνουμε πολλά στον αφορά της ενέργειας και αν κινηθούμε σωστά μπορούμε να δημιουργήσουμε και θέσεις απασχόλησης και να έχουμε βελτίωση της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Σε αυτό το πνεύμα, φέτος, τα βασικά επιτεύγματα των δράσεων μας για το κλίμα ήταν η οθέτηση του οδικού χάρτη για το 2050 προς μια ανταγωνιστική οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και να λαμβάνεται υπόψη στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω η πτυχή του κλίματο. Είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε το δικό χάρτη για το 2050 κατά παρελθόν και δεν θα αναφέρω πολλέ λεπτομέρειε. Εδώ βλέπετε πολύ σαφώ πώ βλέπουμε τι ευφυεί πολιτικέ για το κλίμα, την αποδοτικότητα τη ενέργεια, βελτίωση τη ασφαλού εφοδιασμούς ενέργεια και τα χρησιμοποιήσουμε αυτά σαν κινητήρα για καινοτομία και θέσει απασχόληση. Θεωρούμε ότι είναι ένα σύνολο αυτό και όλο σκοπό των πράξεών μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να μεριμνήσουμε για τη χρήση των σωστών εργαλείων που θα εξυπηρετούν ταυτόχρονα και τους τρεις σκοπούς. Βεβαίως παρακολουθώ μεγάλο ενδιαφέρον τις συζητήσεις σας στα πλαίσια της προετοιμασίας της συνομονωτήσεως του κύριου Πινέδο, κυρίου Πυρίλο και προσβλέπω στην ε, άποψη του Κοινοβουλίου που ελπίζω ότι θα εγκρίνει σαφώ την προσέγγιση. Ο κ. Πυρίλο ζητά περισσότερου πόρου, κυρίω όσον αφορά την αύξηση τη αποδοτικότητα ενέργεια και αυτό μου οδηγεί αμέσω στο επόμενο σημείο μου. Διότι σαν ανακοίνωση για την επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αυξήσει σημαντικά ε, τη συμπερίληψη τη στοιχή του κλίματο του προπολογισμού του Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Είπαμε ότι τουλάχιστον 20% του προπολογισμού κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να υποστηρίξει την προσπάθειά μα για την επίτευξη των στόχων για την καταπολέμηση τη αλλαγή του κλίματο και τι φιλοδοξίε μα. Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει ότι ένα γενικό προπολογισμό που είναι αφορά το κλίμα, αλλά θέλουμε να δούμε τι κάνουμε τι υποδομέ, τι μεταφορέ, την έρευνα, τη γεωργία, την ενέργεια, τι γίνεται και με του άλλου τομεί και πώς όλα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προωθήσουμε ε, την επίτευξη των επιθυμητών στόχων. Νομίζω ότι στείλαμε ένα ισχυρότατο μήνυμα προς τα έξω. Ε, αν θέλουμε να μιλήσουμε για αποδοτικότητα της ενέργειας, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ε, τα ενεργειακά δίκτυα, να έχουμε ευφυεί μετρητές, να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα της ενέργειας στον τομέα της στέγασης. Υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς που μπορούν να δημιουργηθούν θέσει απασχόλησης και μπορούν να δημιουργηθούν γρήγορα και ο οικοδομικός τομέα χρειάζεται ε, την ανάπτυξη και τέτοιου είδους δουλειέ δεν θα μπορέσουν να πάνε στην Κίνα ή αλλού με υπεργολαβία. Να αναφέρω μερικά άλλα πράγματα. Στείλαμε στα κράτη-μέλη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προ ενημέρωση πρόσφατα το μέτρο που εφαρμόζει την οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων που αφορά τη μεθοδολογία για τα αέρια του θερμοκηπίου για τα ορυκτά καύσιμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να αντιμετωπίσει όλα τα καύσιμα που δημιουργούν αέρια του θερμοκηπίου με συνεπή τρόπο, ε, με συγκεκριμένες τιμές και δείκτες συμπεριλαμβανομένων και τιμών για το πετρέλαιο από σχιστόλιθο και από διάφορα ε, αμμόδια δάφη. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η μεθοδολογία που χρησιμοποίησαμε για τα ορυκτά καύσιμα θα είναι παράλληλη με τη μεθοδολογία που ακολουθήσαμε για τα ε, βιοκαύσιμα που ακολουθήσαμε προσέγγιση που αφορά τις διάφορες ζωοτροφές που χρησιμοποιούσαν διαφορετικές τιμές. Όσον αφορά την ποιότητα, την οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων, οι υπηρεσίες μας ολοκληρώνουν τις εργασίες για αξιολόγηση συνεπιών και ετοιμάζουν νομοθετικέ προτάσει. Όσον αφορά τις εκπομπές από έμεση, έμεση αλλαγή της χρήσης της γης μέσω βιοκαυσίμων. Περίπλοκα πράγματα όλα αυτά. Βασικό σκοπός είναι να αποφύγουμε να δημιουργήσουμε μεγάλη βιομηχανία για βιοκαύσιμα και η παραγωγή για βιοκαύσιμα να πάει αντίθετη με την παραγωγή τροφίμων. Είναι πολύ σημαντικό. Η πρόταση αναμενόταν επί μακρόν, χρειαστήκαν περισσότερο χρόνο από ό,τι προβλεπόταν, αλλά θα συμφωνείτε ότι τελικά ε, το σημαντικότερο είναι να πετύχουμε τα σωστά ε, μέτρα, γιατί πολλά δικηβεύονται. Του τελευταίου μήνε προχωρήσαμε πολύ και ελπίζω να μπορέσουμε να θετήσουμε μια πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το τέλο των ενεστώτο έτου. Θα ήθελα να υπογραμμίσω και κάτι άλλο, κυρία Πρόεδρε που σίγουρα θα ενδιαφέρει και την Επιτροπή σας και αυτό είναι το θέμα της συμπερίληψης της των αερομεταφορών ε, στο σύστημα εμπορίου ε, ρήπων της, ε, καταλλαγής ρήπων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Να σας πω ότι σημειώσατε την περασμένη εβδομάδα ότι η ΚΑΟ πήρε μια απόφαση. Είδατε στον τύπο ότι πολλά τρίτα μέρη διαμαρτυρήθηκαν είναι σημαντικό και το Κοινοβούλιο να θυμηθεί ποιο είναι το όλο ιστορικό. Από το 1997 η Ευρώπη προσπάθησε να θεσπίσει νομικά σε διεθνές επίπεδο το θέμα αυτό. Ακόμα εξακολουθούμε να προσπαθούμε. Το 2008 εσείς το Κοινοβούλιο, 27 κράτη-μέλη και η τότε Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίσατε να καλυφθεί και ο τομέας αερομεταφορών μεταφορών στο σύστημα εμπορίου ρήπων και ταιριάζει αυτό με αυτό που έχει αποφασίσει ήδη το ΙΚΑΟ το 2004. Τώρα, σε αντίθεση με το 2004, η Διεθνής ε, Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας είπε ότι λογικό είναι να θέλουμε να ρυθμίσουμε το κλίμα να το κάνουμε μέσω ενός συστήματος εμπορίας εκπομπών και επίσης είναι λογικό να ξεκινήσουμε με ένα περιφερειακό τέτοιο σύστημα. Όταν ε, θεσπίστηκε η σχετική νομοθεσία στην Ευρώπη, φυσικά ήταν σημαντικό να γίνει με τρόπο που δεν θα ε, πλήξει τις ε, ευρωπαϊκές αερογραμμές σε σχέση με τις ανταγωνιστικές άλλες εταιρείε. Οπότε θα πρέπει όλες οι εταιρείες, οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες και οι εξωευρωπαϊκές να τη χάνουν ίση μεταχείριση ό,τι αφορά τις αφήξεις αναχωρήσεις αεροπλάνων. Βέβαια, όταν ε, πρωτοθεσπίστηκε η νομοθεσία αυτή, ε, πολλοί ε, ήταν επιφυλακτική, περίμεναν τις συνέπειες ε, ε, της εφαρμογής της και ε, αναφέρθηκε το θέμα του διαλόγου με τις χώρες που διαμαρτύρονταν κατά του συστήματος, γιατί εμείς έχουμε στην νομοθεσία μας τέτοια διάταξη ότι αν μια τρίτη χώρα εφαρμόζει ισοδύναμα μέτρα, μπορεί να εξαιρεθεί από την εφαρμογή της ε, κοινοτικής νομοθεσίας. Ε, και σε τέτοιες περιπτώσεις έχουμε διάλογο με Ρωσία, Κίνα, Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες και φυσικά αυτή η δραστηριότητα βρίσκεται ε, εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή. Σε ό,τι αφορά την, το προδικαστικό, την προκαταρκτική γνωμοδότηση της 6 Οκτωβρίου σε ό,τι αφορά μια προσφυγή αμερικανικών αερογραμμών. Ε, ήταν σαφής αυτή η προδικαστική απόφαση και λέει ότι όλες οι αξιώσεις ε, των αμερικανικών αεροπορικών εταιριών δεν ευσταθούν και δεν ισχύει ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία είναι κατά της ε, νομοθεσίας UCAT ή κατά του FCCC ή κατά της νομοθεσίας του ICAO ούτε ευσταθεί ότι υπάρχει εξοδοφικότητα. Όλα τα θέματα του προδικαστικού, του προδικαστικού ζητήματος ουσιαστικά έδωσαν δίκιο στην ευρωπαϊκή πλευρά. Βέβαια, πολλές ερωτήσεις θα σας υποβληθούν για το θέμα αυτό. Εμείς συνεχίζουμε τις εργασίες και μερικές φορές χάνουμε την αίσθηση του μέτρου με ε, αυτά που διαβάζουμε στον ε, τύπο. Φαίνεται ότι ότι θα αυξηθούν τα ε, ευρωπαϊκά εισιτήρια και θα πολλαπλασιαστούν οι τιμές των εισιτηρίων ε, Ευρώπης-Αμερικής. Εδώ μιλάμε για αύξηση του το 10 ευρώ, αλλά το 85% το πρώτο χρόνο, το 82% τα επόμενα χρόνια ε, που θα δοθούν δωρεάν στις αεροπορικές εταιρείες και όχι τα 50 ευρώ αύξηση που ακούστηκε, διαβάσαμε στον τύπο. Οπότε Μία πτήση Λονδίνο-Νέα Υόρκ θα είναι 1,5 ευρώ η επιβάρηση. Φραγκφούρτη-Πεκίνο θα είναι γύρω στα 2 ευρώ η επιβάρηση. Φαντάζομαι συμφωνείτε κι εσείς ότι πολύ δύσκολα θα βρούμε κάποιο που θα θέλει να σταματήσει στο Αμπουνταβί το Ντουμπάι, μόνο και μόνο για να εξοικονομήσει 2 ευρώ, αν μπορεί να έχει απευθείας πτήση Ευρώπη-Πεκίνο θα προτιμήσουν ε, να μην κάνουν διάμεση στάση ε, και να, για να εξοικονομήσουν μόνο και μόνο τα 2 ευρώ. Για να μην ξεχνούμε πόσο επιπλέον καύσιμα θα χρειαστεί μια τέτοια στάση. Κύριε Πρόεδρε, να αναφερθώ στις βασικές μας προτεραιότητες για το 2012 και το πρόγραμμα δράσης. Καταρχήν θέλουμε καιρό να εφαρμόσουμε το πακέτο για την ενέργεια και το κλίμα. Πρωταρχική προτεραιότητα. Ε, εν ώψη και τη τρίτη φάση του EU του Συστήματος Εμπορία Εκπομπών που θα ξεκινήσει το 2013. Επίση, ε, ετοιμάζουμε κάποιε πρωτοβουλίε ε, για τι κλιματικέ αλλαγέ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Περιμένουμε αναθεώρηση του κανονισμού για το, διο... για το διοξείδιο του άνθρακα για φορτηγά και αυτοκίνητα. θα επιτρέψουμε μείωση των εκπομπών με τον κανονισμό αυτό και επίση ενίσχυση τη ε, καινοτομίας. Ό,τι αφορά τις εκπομπέ, τη θαλάσσιε μεταφορέ. θέλουμε σφαιρική η παγκόσμια δράση. Και αν δεν υπάρξει μέχρι τέλη του έτους κάποια ε, παγκόσμια πρωτοβουλία, θα ε, προετοιμάσουμε μια κοινοτική προσέγγιση. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες εδώ, θα επανέλθουμε στο θέμα. Να σας ενημερώσω ότι ο Επίτροπος Κάλλας, Επίτροπος Μεταφορών και εγώ το τελευταίο χρόνο είχαμε ένα φόρουμ των ενδιαφερομένων μερών, συναντήσεις με πολλούς ενδιαφερόμενους και εκπροσώπους του κλάδου προκειμένου να εξετάσουμε το κατά πόσο θα πρέπει να τηρήσουμε αυτή τη ε, δέσμευση που μας ενέθεσε το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και με ποιο τρόπο θα πρέπει να γίνει. Οπότε ήδη συμπεριλαμβάνουμε συζητήσεις στους ενδιαφερόμενους και για το χρόνο θα αναθεωρήσουμε την ε, νομοθεσία για το ΕΦΚΑΣ με βάση την πρόσφατη ε, έκθεση που μιλάει για την ανάγκη αποτελεσματικής μείωσης και επικερδούς των εκπομπών. Επίσης θα πρέπει να ενεργοποιηθούμε δραστήρια στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για τη μείωση των κλιματικών αλλαγών, αλλά θα εξαρτηθεί αυτό και από την έκβαση του Ντέρμπαν. Και ε, με τον Ντέρμπαν θα τελειώσω κύριε Πρόεδρε. Θα μπορούσα να μακρηγορήσω, αλλά προτιμώ να είμαι λακωνική. Ε, στο Ντέρμπαν έχουμε να αντιμετωπίσουμε κυρίως τρία θέματα. Πώς εφαρμόσουμε όλα όσα έμειναν εκκρεμή και δεν συμφωνήθηκαν στο Κανκούν Μπορεί να ακούγεται βαρετό αυτό για τους πολιτικούς, αλλά υπάρχει ένας μακροσκελής κατάλογος θεμάτων που πρέπει να εφαρμόσουν. Δεν αρκεί να λαμβάνονται αποφάσεις, δεν αρκεί να αποτυπώνεται μια απόφαση στο χαρτί. Υπάρχουν πολλά θέματα. Επιστημονική τεχνολογική επιτροπή, χρηματοδότηση υποδομών, δρόμων, αλλαγή χρήση γη κτλ. Πολλά ζητήματα συναφή που θα πρέπει να διευθετηθούν και εκεί περιμένουμε πρόοδο στον Τέρμπαν. Ε, ορισμένα ζητήματα δεν αναφέρθηκαν καν στο Κανκούν. Αναφέρθηκε η πολιτική αεροπορία, ναυτιλία, ε, μηχανισμοί που θα προσανατολίζονται στην αγορά, ε, μηχανισμός καθαρής ανάπτυξης, καλύτερη κατανομή των προϊόντων, ε, να, μην ξεχνούμε τους ε, πιο ευάλωτους, τις πιο προβληματικές χώρες, να έχουμε μακροπρόθεσμα σχέδια. Υπάρχει ένα, ένας μεγάλος κατάλογος τέτοιων θεμάτων που θα πρέπει να συζητηθούν στον Τέρμπαν. Επίσης υπάρχει και το θέμα της δεύτερης περίοδου δέσμευσης για το πρωτόκολλο του Κιώτο. Θα διαβάσετε πολλά στον τύπο για το θέμα αυτό μετά την έναρξη της διάσκεψης. Φυσικά αναφέρθηκε η πρόταση να αναλυθεί από την Ευρώπη δεύτερη περίοδο δέσμευση για το πρωτόκολλο του Κιώτο. Βρισκόμαστε στα τέλη του πρώτου χρόνου που ε, εκπνέει η πρώτη περίοδο δέσμευση. Όχι η ίδια η σύμβαση, αλλά η πρώτη περίοδο δέσμευση τη σύμβαση εκπνέει. Είπαμε λοιπόν το εξή. Ναι, μεν η Ευρώπη είναι διατεθειμένη, είναι πρόθυμη να ε, ενταχθεί σε μια δεύτερη περίοδο δέσμευση, παρόλο που ξέρουμε ότι η Ρωσία, ο Καναδά και η Ιαπωνία τελικά δεν θα δεχτούν μια δεύτερη περίοδο δέσμευσης, αλλά είπαμε επίσης ρητά και κατηγορηματικά ότι κάτι τέτοιο θα γίνει υπό όρου και όχι ανεπιφύλακτα, υπό όρου που θα λαμβάνουν υπόψη ε, την, το περιβαλλοντικό παράγοντα και υπό τον όρο ότι και άλλοι σημαντικοί οικονομικοί εταίροι, άλλες σημαντικέ οικονομίε θα μας πούν πότε εκείνε σκοπεύουν να αναλάβουν αντίστοιχες προσπάθειες. Τι σημαίνει αυτό σημαίνει ότι φυσικά δεν μπορούμε να έχουμε την νομικά δεσμευτική συμφωνία που επιθυμούσαμε εμείς, που θέλουν και οι επιχειρηματικοί μα κύκλοι. Αυτό αποκλείεται στον τέρμα, να έχουμε νομικά δεσμευτική συμφωνία. Βλέπετε τι συμβαίνει στη ΣΥΠΑ, βλέπετε τι συμβαίνει και αλλού στον κόσμο. Αλλά τι η Ευρώπη να χτίζει γέφυρες ε, και να μπαίνει σε δεύτερη περίοδο δέσμευσης μόνη της όταν δεν ακολουθεί κανένα σε αυτό τον δρόμο. Γι' αυτό είπαμε ότι θα πρέπει τουλάχιστον να καταρτήσουμε ένα νοδικό χάρτη στο Ντέρμπαν με σαφές χρονοδιάγραμμα. Γιατί είμαστε όλοι μεγάλες οικονομίες. Βραζιλία, Ήπα, Κίνα. Αυτές οι οικονομίες θα πρέπει αυτές οι χώρες να μας πούν πότε σκοπεύουν να ενταχθούν σε αυτή τη δέσμευση. Και τέλος, ξέρετε ότι σήμερα έχουμε δύο κατευθύνσεις, δύο μπλοκ. Οι αναπτυσσόμενες χώρες από τη μια πλευρά που δεν έχουν καθόλου δεσμεύσεις, καθόλου υποχρεώσεις από το Κιώτο, όλα προαιρετικά σε προαιρετική βάση οικειοθελώς, ενώ οι αναπτυγμένες χώρες είναι υποχρεωμένες να έχουν συγκεκριμένες επιδόσεις. Πιστεύω ότι τον 21ο αιώνα ε, δεν θα πρέπει να συνεχιστεί για πολύ αυτός ο διαχωρισμός μεταξύ αναπτυσσομένων και αναπτυγμένων χωρών. Η Κίνα δηλαδή είναι αναπτυσσόμενη χώρα όπως το Μαλί και το Μαλάουι. Είναι σαφές ότι ο κόσμος θα πρέπει να χαρακτηριστεί βέβαια από διαφορετικέ δεσμεύσει και σίγουρα οι ανεπτυγμένε χώρε θα πρέπει να αναλάβουν δεσμεύσει πιο φιλόδοξε και πιο γρήγορα από τι αναπτυσσόμενε χώρε. Αλλά να ισχύει η ίδια νομική δέσμευση. Νομίζω ότι αυτό είναι από τα σημαντικά θέματα που θα εξεταστούν στο Τέρμπαν. Οπότε φαντάζεστε η συζήτηση δεν θα είναι καθόλου εύκολη, αλλά φαντάζομαι πως θα συμφωνείτε μαζί μου ότι είναι επιτακτική ανάγκη στις αρχές του 21ου αιώνα να συμφωνήσουμε ότι είμαστε αλληλοεξαρτούμενοι ε, και δεν μπορούμε να έχουμε ε, δύο μέτρα και δύο σταθμά και μόνο λίγες χώρες να φέρουν ε, το νομικό βάρος και τη νομική υποχρέωση για μέτρα. Ε, ακούσαμε ότι καμία, ε, ότι οι χώρες που δεν είναι στο ΩΣΑ αυτή τη στιγμή ε, ε, το 70% είναι επίθεση για το 70% της αύξησης ε, ενέργεια, κατανάλωσης ενέργειας. Αν συνεχίσουμε αυτή την πορεία χωρίς δεσμεύσει εκ μέρους τους, δεν θα πρόκειται να τηρήσουμε το, στόχο για τη μία αύξηση κατά δύο βαθμούς Κελσίου. Πιστεύω ότι στον Τέρμα θα πρέπει να ορίσουμε ένα πιο δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για να ξέρουμε πότε οι εταίροι μας θα εστερνιστούν αυτές τις δεσμεύσεις. Και το, το θέμα της χρηματοδότησης, ε, εξίσου σημαντικό. Εμείς α, ε, ε, τηρούμε τις υποχρεώσεις της Κοπεχάγης δεν θα πρέπει λοιπόν η μόνη έκβαση του Ντέρμπαν να είναι λύση της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης και να μείνουν όλα τα υπόλοιπα θέματα εκρέμη. Θέλουμε συνολικό πακέτο και δεν πρόκειται να χρηματοδοτήσουμε κάτι αν δεν γίνονται ε, σαφείς προσπάθειες σε συγκεκριμένους τομείς και θέλουμε ισορροπημένο πακέτο. Αυτά έτσι έχουν τα πράγματα τρει εβδομάδες πριν τα εγγένεια της διάσκεψης του Ντέρμπαν. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα, αλλά από την πρόσφατη εμπειρία μου μπορώ να σας πω ότι πολλέ χώρες αρχίζουν και συντάσσονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιλαμβάνονται ότι αν εμείς μπούμε μόνοι μας στην δεύτερη περίοδο δέσμευση σαν θα είναι πολύ δύσκολο να χαρακτηρίσουμε επιτυχία για το περιβάλλον των Ντέρμπαν, Γιατί δεν θα έχουμε επιπλέον μείωση του διοξιδίου του άνθρακα. Αν θέλουμε μείωση του διοξιδίου του άνθρακα, θέλουμε δεσμεύσει και από άλλου εταίρου. Περί αυτού πρόκειται. Αυτό θα είναι το διακύβευμα του Ντέρμπαν. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Επίτροπε. για τις ε, εξηγήσει για το τι σημαίνει αυτή τη στιγμή και τι μας περιμένει. Προσεχώς, αν μου επιτρέπετε, θα ξεκινήσω αμέσως με τους συναδέλφους. Πρώτα απ' όλα να ακούσουμε τον... την κυρία Γιόρταν Σίσελη. να έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Χέντεγκάρντ. Πάντα βεβαίως είστε ανοιχτοί για να συζητήσετε μαζί μας και στην Επιτροπή Βιομηχανίας και Περιβάλλοντος. Έχω κάποια σχόλια. Αναφέρατε τον οδικό χάρτη 2050 που θα υιοθετηθεί του χρόνου. Ελπίζω η ατμόσφαιρα στο Συμβούλιο να γίνει πιο θετική. Και ε, ε, το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την οικονομία και είναι κατ' ουσίαν ένας οδικός χάρτης της φιλοδοξίας μας αλλά συνεισφέρει και στην σταθερότητα. Οπότε το ερώτημά μου είναι το εξής. Σύμφωνα με την άποψή σας λοιπόν, όχι επίσημη θέση, άποψη, εάν ο δικός αυτός χάρτης υιοθετηθεί, τι θα πρέπει να αλλάξουμε μέχρι το 2020. Στην πρώτη μου ερώτηση. Δεύτερον, αναφέρατε τον προϋπολογισμό και πως 20% του προϋπολογισμού πρέπει να πάει στο κλίμα. Ακόμη περισσότερα θεωρώ εγώ εάν είναι να είμαστε σοβαροί, γιατί εδώ πέρα τη γεωργία, διαρθρωτικά ταμεία, ανάπτυξη κτλ. Οπότε, θα ήθελα εγώ να επισημάνω το εξή. Ο προπολογισμό τη Ένωση κατά βάση στηρίζει μεγάλα έργα. Όμω, όταν μιλάμε για την κλιματική αλλαγή, να ξέρουμε πως είναι σημαντικά τα μικρά έργα. Οπότε εγώ κάνω την εξή έκκληση αυτά τα οποία αναφέρονται ως κλιματική αλλαγή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τα απαραίτητα έργα, όχι μόνο τα μεγάλα έργα, αλλά και τα μικρά. Τρίτον, το Ντέρμπαν. ορίζω την προσέγγισή σας. Θεωρώ πως χρειάζεται μια ρεαλιστική προσέγγιση και αν ε, κάνει τα πράγματα η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως είπατε, αυτό θα είναι κάτι το θετικό. Έχω ένα ερώτημα όσον αφορά το Κιώτο 2. Είπατε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ναι, αλλά υπό όρους και οι όροι αυτοί είναι οι άλλες μεγάλες οικονομίες να συμφωνήσουν και εκείνες, να συστρατευτούν μαζί μας. Θα ήθελα να γνωρίζω το εξής. Με ποιο τρόπο και πότε θα πρέπει να γίνουν αυτές οι δεσμεύσεις. Σύμφωνα με τους ειδικού, θα πρέπει να μειώσουμε τις κομπές διοξιδίου του άνθρακα μέχρι το 2015 το αργότερο και είναι εξαιρετικά σημαντικό να υλοποιηθεί ένας τεχνολογικός μηχανισμός. Εδώ πέρα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να εφαρμοστεί αμέσως η αρχή του να χρησιμοποιούμε την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχουμε ήδη την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία, οπότε δεν χρειάζεται να περιμένουμε στο μέλλον. Οπότε μια συμφωνία για τη μεταφορά της τεχνολογίας είναι σημαντική. Θεωρώ πως αυτό είναι προτεραιότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε για τη διεξοδική σας ε, παρουσίαση και ομιλία. Um, Όλοι μιλούμε για καινοτομία αυτές τις μέρες. Όμως τι βλέπω εγώ είναι πολύ δύσκολο να το πετύχουμε ε, σαν στόχο την καινοτομία. Γλιστράει σαν σαπούνι. Προσπαθούμε να πλύνουμε τα χέρια μας, μας φεύγει το σαπούνι από τα χέρια. Έτσι τα βλέπω εγώ. Και όλα τα προγράμματα και τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βλέπω ότι υπάρχει μια τάση προς την έρευνα. Δεν βλέπω όμως ε, να υπάρχει ε, αρκετή έφεση προς την καινοτομία. Χρησιμοποιείται αυτή η λέξη, αλλά στην πράξη δεν το βλέπω. Ε, Αν μιλάμε καινοτομία προς ποια κατεύθυνση. Αυτά σαν γενικά σχόλια. Μιλάμε για πράσινη ανάπτυξη. Το επίθετο πράσινο πιέζεται λόγω της οικονομικής κρίσης. Το πράσινο πώς θα το προωθήσουμε στο πράσινη ανάπτυξη, διότι πολλές επενδύσεις εξακολουθούν να πηγαίνουν στην άλλη κατεύθυνση. Είπατε ότι η ανάπτυξη πρέπει να συνδέεται με την απασχόληση και δεν θέλουμε οι θέσει απασχόληση να πάνε στην Κίνα. Όμως οδηγίες όπως η έκθεση ΡΟΣ του περασμένου χρόνου είδαμε ότι δεν τροποποιήθηκε ούτως ώστε ε, ε, ε, να απαγορευτούν οι ηλιοσυλλέκτες ε, που χρησιμοποιούν υλικά τοξικά από την Κίνα. Υπάρχουν σε άλλες αγορές ε, πιο βιώσιμα προϊόντα και αυτό πρέπει να το προσέχουμε από πού ε, χρησιμοποιούμε τα προϊόντα. Πρέπει σε όλες τις οδηγίες να υπάρχει αυτός ο έλεγχος. Το μέτρο αυτό ε, οδηγεί, το μέτρο που είναι φιλικό προς το περιβάλλον ε, δημιουργεί θέσεις απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι φιλικό προς το περιβάλλον αλλά δεν δημιουργεί θέσεις απασχόλησης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε μια νέα διάσταση στον αυτό το κλίμα, η αποδοτική χρήση των πρώτων υλών. Μας τελειώνει η φυσική πόρη και αυτό είναι κάτι που όλο και πιο πολύ προσέχετε και τονίζετε. Εσείς προφανώς δίνεται μεγάλη προσοχή στην εκπομπή διοξιδίου του άνθρακος. Πού ταιριάζει αυτό με την αποδοτικότητα των πόρων, με το ρίο συν 20 του επόμενου χρόνου. Δεν θέλουμε να έχουμε τεχνολογία που είναι φιλική όσον αφορά το περιβάλλον και φιλικά όσον αφορά το διοξίδιο του άνθρακος, αλλά θέλουμε να υπάρχει και φιλικότητα των προϊόντων και των μηχανημάτων έναντι των πρώτων υλών. Τώρα η των πόρων. Είναι σημαντικό το, θέμα. Μπορεί να δώσει πολλές θέσεις απασχόλησης και πολλά ωφέλιμα αποτελέσματα στον φάτο το του άνθρακος. Θέλουμε η οδηγία για την αποδοτικότητα της ενέργειας να επεκταθεί και προς τις ε, ιδιωτικές ε, κατοικίες, ε, τις εργατικές κατοικίες. Ε, αν θέλουμε να είμαστε αποδοτικοί, να καλύψουμε το βρύτερο δυνατό πεδίο όλα τα κτίρια. Και όχι μόνο αυτά τα κτίρια που ελέγχουμε άμεσα. Ε, αερομεταφορές. Συμφωνώ μαζί σας. Πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι. Χρειάστηκε χρόνος. Ξεκίνησε εδώ και πολλά χρόνια άλλη προσπάθεια. Πρέπει να ηγηθούμε. Όμως, έχω την Κοπενχάγη στο μυαλό μου, όπως και εσείς. Μου κόλλησε η Κοπενχάγη. Αυτά που συνέβησαν. Ήμασταν πολύ φιλόδοξοι, ήμασταν πολύ γενναίοι δεν καταφέραμε όμως να πείσουμε και τους άλλους. Και αυτό φοβάμαι ότι θα συμβεί και με το θέμα της εμπορίας ρήπων στη δομέα της αερο... των αερομεταφορών. Φοβούμε τα αντίπεινα, το φοβούμε. Αν καθυστερήσουμε, αν αργήσουμε, τι θα γίνει. Υπάρχει οικονομική κρίση. Εταιρείες που θα χρεοκοπήσουν. Ίσως κερδίσουμε στο τέλος είπα και εκείνα, να έρθουν μαζί μας, αλλά ίσως να γίνει πολύ αργά. Να είναι επίρρεια νίκη και να εξαγοραστούν από τους Κινέζους οι εταιρείε μας. Αν θέλουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε το θέμα των αερομεταφορών, γιατί να μην αλλάξουμε και τους κανόνες για το ΦΠΑ. Να, λήξει, να λήξουν οι εξαιρέσει και όλα τα προνόμια που έχουμε δώσει στον τομέα. Τέλος, το Ντέρμπαν, Εξίσου σημαντικό θέμα. Ε, συμφωνώ μαζί σας απόλυτα ότι είναι πολύ σημαντική η υλοποίηση όλων αυτών. Σημαντικό να έχει κανείς καλά σχέδια, σημαντικότερο, πολύ σημαντικότερο να τα υλοποιούμε βάσει του σχεδίου μας. Όλοι προσπαθούμε να πετύχουμε συμφωνία στο Ντέρμπαν. Δεν τα καταφέραμε στην Κοπενχάγη, πετύχαμε εν μέρη το στόχο μας στο Κανκούν. Μήπως θα ήταν καλύτερο στο μέλλον να προσπαθούμε μικρές μερικές συμφωνίες που μας οδηγούν στον τελικό μας στόχο. Ευχαριστώ και καλή τύχη. Η κυρία Χολ. Ναι, ευχαριστώ κυρία Επιτροπέ για την αναλυτική σας παρουσίαση που βεβαίως όπως πάντα μας βοηθάει. Υπήρχαν ε, κάποια θέματα στα οποία θα ήθελα να ζητήσω περισσότερες λεπτομέρειες. Με ενδιαφέρει αυτό το οποίο είπατε για την οδηγία ποιότητας καυσίμων και σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Ζητήσα, συναντήσατε ευρωβουλευτές αρκετές, σε αρκετές περιπτώσεις. Ενδιαφέρον ήταν το ότι τονίσατε το ότι θα υπάρξουν συγκεκριμένες τιμές για όλα τα καύσιμα και είπατε πως υπάρχει ένας παραλληλισμός μεταξύ των όσων ζητάμε από τα ορυκτά καύσιμα και τα βιοκαύσιμα. Και ήθελα να σας ρωτήσω κάποια πράγματα παραπάνω σε σχέση με την έμεση αλλαγή χρήσης γης. Γιατί ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα, ακούμε φήμες για το τι ακριβώς θα προτείνει η Κομισιόν επ' αυτού και για το εάν θα έχουμε ξεχωριστές τιμές για κάθε ζωοτροφή, βιοκαύσιμο και αν θα προκύψουν αμέσως ή μετά από λίγο χρόνο. Το γενικότερο μου ερώτημα, εν πάση περιπτώσει, είναι αυτή τη στιγμή επεξεργάζεστε κάποιου είδους εξορθολογισμό η σχέση μεταξύ της αλλαγής χρήσης γης και της ποιότητας καυσίμων επισήμως ή ανεπισήμως. Το δεύτερο μου ερώτημα αφορούσε τον Τέρμπαν. Αναφέρατε το μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και το πώς δεν ε, μπόρεσε να ε, δημιουργήσει έργα ε, ειδικά στις χώρες της υποσαχαρίου Αφρικής. Και αναρωτιέμαι πώς συνεννοείστε με τον Επίτροπο Πίμπαλξ και τις προσπάθειες που καταβάλει για πρόσβαση στην ενέργεια από όλους και με ποιο τρόπο μπορούμε να κάνουμε το μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης να επιτύχει αυτούς τους στόχους για πρόσβαση στην ενέργεια. Ευχαριστώ. Η κυρία Καρβάλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την Επίτροπο για τις ευαίσθητες όπως πάντα εξήγησει για το μελλοντικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις προσδοκίες μας ε, από τη διάσκεψη του Ντέρμπαν. Έχω μία ερώτηση σχετική με το Τέρμπαν και τη δεύτερη περίοδο δεσμεύσεων. Γιατί φαντάζομαι θα είναι δύσκολη η απόφαση που θα κλείθει να λάβει η Ευρώπη. Μίλησατε για όρους. Ερωτώ λοιπόν. Δεν είναι σκόπιμο να προσθέσουμε και νέους δύο όρους. Φαντάζομαι θα το έχετε σκεφτεί. Θα θέλαμε να μας πείτε ποιους ακριβώς όρους συγκεκριμένα έχετε υπόψη όταν λέτε ότι υπό όρους θα πρέπει να ε, περάσουμε στη δεύτερη περίοδο δεσμεύσεων. Κατά τη γνώμη μου, ο όρος θα ήταν ε, ο τρόπος αντιμετώπισης του θέματος διαρροής άνθρακα και των ενεργειοβόρων ε, βιομηχανικών κλάδων. Δηλαδή, μπορούμε να συνδυάσουμε την αντιμετώπιση αυτών των ενεργειοβόρων ε, κλάδων με δεσμευτικούς ε, στόχους για την οικονομία. Δηλαδή να έχουμε κάποιες κλαδικές τομεακές συμφωνίες για συγκεκριμένους ε, κλάδους και να το συνδυάσουμε με συγκεκριμένη αντιμετώπιση του στα πλαίσια του πρωτοκόλλου του Κιώτο. Έχουμε ήδη ένα κατάλογο υποχρεώσεων έχουμε συγκεκριμένους οικονομικούς παγκόσμιους στόχους και έχουμε, να έχουμε και γενικούς στόχους για συγκεκριμένους τομείς. Περίπου δηλαδή αυτό που κάνετε για την αεροπορία ή ε, και μέχρι σε ενός βαθμού και για τα δάση. Δηλαδή, να λάβετε υπόψη και την ανταγωνιστικότητα, το πιθανότητα πλήξης της ανταγωνιστικότητας, πλήγματος της ανταγωνιστικότητας για ορισμένους ευρωπαϊκούς κλάδους κατά τη δεύτερη περίοδο δέσμευση. Το σκέφτεστε, το έχετε υπόψη ήδη αυτό, θα το λάβετε ε, υπόψη της διαπραγματεύσεις. Σε ό,τι αφορά το CDM, θα γίνει ένας ανασχεδιασμός του CDM των στόχων της χιλιετίας, των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. Ούτε μείωση των τιμών έχουμε, ούτε, βελ, ούτε βελτίωση κατάστασης ή βοήθεια των πιο ευάλωτων πληθυσμών στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Ε, χωλένουμε πολύ, στερούμε πολύ σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ίδια τη σύμβαση, θα θέσετε ως όρο για τη δεύτερη περίοδο τη δεσμεύσεων τον ανασχεδιασμό των ε, αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. Ε, συγγνώμη για το μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης, γιατί αν ε, δεν λάβουμε υπόψη και τους δύο στόχους, είναι πολύ δύσκολο να βρούμε ισορροπημένη λύση. Ποια είναι η γνώμη σας για τους δύο αυτούς στόχους, για το μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης. Και... Ευχαριστώ, θέλω και εγώ να κάνω ένα ερώτημα. Και σε πολλά και εντός και εκτός του Κοινοβουλίου Ακούγεται η άποψη πως ε, θα πρέπει να συνεργαστούμε τις λιγότερο ανεπτυγμένες ε, χώρες ε, για το διοξείδιο του άνθρακα. Δεν το κατάλαβα αυτό, δεν το έχω καταλάβει ακριβώς γιατί με τις λιγότερο αναπτυγμένες. Εντάξει, οι, αυτές που είναι σε πορεία ανάπτυξης ε, και έχουν την δυναμικότητα, ναι, το καταλαβαίνω, αλλά τι να συνεννοηθούμε με τον Μπουρούντι και το Μαλί όταν ε, μιλάμε κατ' ουσίαν για Ρωσία, Ινδία, Βραζιλία. Ίσως να μην έχω καταλάβει καλά. Θα ήθελα μία εξήγηση. Ευχαριστώ. Ωραία. Οπότε θα σταματήσουμε εδώ πέρα και θα δώσουμε στην κυρία Επίτροπο την ευκαιρία να απαντήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σίσλεη, για τον οδικό χάρτη. Τι θα αλλάξει με την υιοθέτηση του οδικού χάρτη. Με βάση τον οδικό χάρτη θα δοθεί η έμφαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Αυτό θα αλλάξει ό,τι φορά ε, το 2020. Επίσης, θα πρέπει να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας στην Ευρώπη για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Γι' αυτό συνδέω με το, το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, το πακέτο για τις υποδομές, τα διαρθρωτικά ταμεία, προκειμένου να προωθήσουμε τους στόχους μας για την ενεργειακή αποδοτικότητα, που είναι ένας από τους στόχους ε, για τα 3.20 και, το, και τη στρατηγική του 2020. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στην Ευρώπη. Εκεί θα δούμε πραγματικά τη διαφορά. Και βλέπουμε και τη συνέπειες ε, του δικού χάρτη για λιγότερο, ε, λιγότερη χρήση άνθρακα. Και οι, ε, διάφορες, οι διάφοροι, βιομηχανικοί, οι διάφοροι βιομηχανικοί κλάδοι έχουν το δικό τους οδικό χάρτη. Και την επόμενη εβδομάδα θα δούμε και μια νέα βιομηχανία που θα υποβάλει το δικό τη οδικό χάρτη. Βλέπετε ότι αντίστοιχε προσπάθειε γίνονται σε διάφορου βιομηχανικού κλάδου και είναι πολύ θετικό αυτό. Επίση ε, και στι πολιτικέ των μεταφορών. Όχι μόνο η Επιτροπή ε, και για τον προπολογισμό, αλλά και οι χώρε ε, και οι δήμοι και οι κοινότητε στον προγραμματισμό του αρχίζουν και λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη μείωσης για το 2050 αλλά και τα προηγούμενα ορόσημα το 2030 και το 2040 και τα λαμβάνουν αυτά υπόψη στον προγραμματισμό των κλαδικών τους πολιτικών. Σε ό,τι αφορά την, το πρασίνισμα της ΚΑΠ και αυτό είναι πολύ σημαντικό και λαμβάνεται υπόψη. Θέλουμε γενικώ μια πιο πράσινη ανάπτυξη σε ό,τι αφορά τα μεγαλεπίβολα σχέδια, θέλουμε τέτοια μεγάλα, μεγάλης εμβέλεια σχέδια. Τώρα, ως προς τον προϋπολογισμό, θα οριστικοποιήσουμε την πρότασή μας μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Προβλέπεται σημαντική αύξηση του τμήματος του Life Plus που αφορά το περιβάλλον. Και αυτό προκειμένου να ενισχύσουμε και κάποια μικρά προγράμματα που είναι ε, καλά, αλλά χρειαζόμαστε μεγάλες ευέλειες προγράμματα για να είναι πιο σημαντικός ο αντίκτυπος. Επίσης, ε, κυρία Μάκης, μιλήσατε για αυτό το, την καινοτομία. Ε, έχουμε ένα καλό παράδειγμα. Έχουμε 300 εκατομμύρια άδειες που θα μπουν σε πληστηριασμό, θα δημοπρατηθούν, κάτι που θα δώσει έναυσμα για τις νέες τεχνολογίες ανανεώσιμων και ε, δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα. Επίσης και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέχρι ε, την 9η ε, Φεβρουαρίου θα ιεραρχήσουν τα διάφορα σχέδια που έλαβαν από τα κράτη-μέλη και του χρόνου του 2012 θα δούμε ποια σχέδια θα προωθηθούν και θα εγκαινιαστούν. Έτσι μπορούμε να είμαστε πολύ πιο συγκεκριμένοι, γιατί δεν είναι να αναμασάμε συνέχεια τον όρο ε, καινοτομία και να τον έχουμε μαϊδανό, αλλά να αποτυπώνεται στην πράξη συγκεκριμένα σχέδια. Επίσης, ε, με ρωτήσατε και εσείς κύριε Καρβάλη και κύριε Σιζηλέ ποιοι είναι οι όροι που θα διαπραγματευτούμε για να μπούμε στη δεύτερη περίοδο δεσμεύσεων στον Τέρμπαν. Και άλλοι σημαντική εταίροι μας ε, έχουν σημαντική εκπομπή και είναι σημαντικέ οικονομίε. Θέλουμε έναν χρονικό ορίζοντα, το 2015 για παράδειγμα, και μέχρι τότε να ολοκληρώσουμε τι λεπτομεριακέ συμφωνίε για το από πότε θα μπουν στη δεύτερη περίοδο δεσμεύσεων, το 2020 για παράδειγμα, για να είμαστε βέβαιοι ότι και για αυτού θα ισχύσουν, αν όχι οι νέοι στόχοι και οι νέε υποχρεώσει, τουλάχιστον ό,τι και αν αποφασίσουν να κάνουν να έχει να έχει την ίδια νομική αξία, την ίδια νομική ισχύ. Αυτό προσπαθούμε να εξηγήσουμε. Και θα έχουμε και άλλους ώρες για το EUCF και το θέμα της, ε, της ε, περιβαλλοντικής ακαιρεότητας του παρόντος συστήματος. Και εκεί θα πρέπει να σημειωθεί πρόοδος. Και όλα αυτά δεν είναι απλές προθέσεις, αγαθές προθέσεις, ότι κάποια στιγμή γενικά και όριστα στο μέλλον κάποιο θα μας ακολουθήσει. Θέλουμε συγκεκριμένα βήματα σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Και κάτι άλλο. Αυτή δεν είναι, αυτό δεν είναι το ιδανικό, το ιδεώδης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς ήμασταν πολύ πιο φιλόδοξοι και περιλα, περιμέναμε πολλά χρόνια για να μπούμε στη δεύτερη περίοδο δέσμευση. Αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι είναι εφικτό για τις υπόλοιπες μεγάλες οικονομίες. Την Κίνα, τη Ρωσία, τη ΣΥΠΑ και να φροντίσουμε να καταρτιστεί και ο δικός χάρτης. Διαπιστώνουμε τι δυσκολίες ε, περιέχει όλη η διαδικασία. Και δυστυχώς δεν έχουμε αρκετό χρόνο. Πρέπει να δείξουμε μια φιλοδοξία και ήδη πολύ χρόνο, αλλά είναι η μόνη μας ευκαιρία. Και εντάξει, μπορούμε να λέμε κρίμα, καθυστερούμε, οι άλλοι δεν μας ακολουθούν, αλλά το θέμα είναι να μην χάσουμε τα κεκτημένα των προηγούμενων χρόνων, ούτε και αυτό μας ενδιαφέρει. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν ε, να κρατήσουμε την πορεία μας σταθερή, λογικά. Γιατί δεν έχει νόημα να λέμε εμείς ναι και οι άλλοι, ε, η Νέα Ζηλανδία, άλλες χώρες να λένε όχι. Κυρία Μέρκης, είπατε που έγινε η συνέργεια μεταξύ της ενεργειακής αποδοτικότητας, της αζεντέντας για το 2020 ε, και το περιβάλλον. Φυσικά υπάρχει συντονισμός μεταξύ των ε, χαρτοφυλακίων των επιτρόπων. Και βλέπουμε την οδηγία για τη φορολογία ή την ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης. Βλέπουμε πώς προσπαθούμε τη φορολογία να την προσανατολίσουμε στις, στους πόρους και την ενέργεια και να την αποδεσμεύσουμε κάπως από τους μισθούς. Έτσι νομίζω θα έχουμε μια πιο ολιστική αντιμετώπιση της ενέργειας και του κλίματος. Σε ό,τι αφορά το γύρο Euro Plus ε, και τις προσπάθειές μας για την Αφρική, πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε ως προτεραιότητα στην Ευρώπη να εξασφαλίσουμε πρόσβαση σε Φόρο βιώσιμη ενέργεια. Και μια τέτοια διάσκεψη μπορεί να είναι τα πάντα και τίποτα και να καταλήξουμε σε ένα δέντρο, σε ένα μακροσκελές ευχολόγιο και σε καμία αυτή ενέργεια. Νομίζω ότι η πρόσβαση σε βιώσιμη ενέργεια θα είναι κεντρικό σημείο. Και αυτό θα είναι, αυτός είναι και ο στόχος μας. Ε, άλλωστε αυτό ζήτησε και το πάνελ του ΟΗΕ του Μπανκιμούν, μια τέτοια σύσταση και ελπίζω να ληφθεί υπόψη όντω ε, και να είναι μία από τις συστάσεις του Ντέρμπαν. Ε, για την, ε, τσαρομεταφορέ, η κυρία Μάκη είπε ότι φοβάται αντίπεινα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία φτιάχτηκε με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να αποφεύγει ακριβώς ανταγωνιστικό μειονέκτημα να δημιουργείται για τις ευρωπαϊκές εταιρείε. Αυτοί που διαμαρτύρονται κατά της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, τι θέλουν να κάνουν. Κάντε αυτό που θέλετε για την Ευρώπη και μόνο. Κάντε ό,τι θέλετε στην Ευρώπη. Αλλά σας παρακαλώ μην πειράσετε τις δικές μας αεροπορικές εταιρείε. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε πολύ μειονεκτική θέση για τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείε. Αν το κάναμε μόνο για τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο θα ήταν και παράξενη λύση. θα βλέπατε πολλές δημιουργικές διαδρομές. Θα κάνανε κύκλους για να αποφύγουν να πετάξουν πάνω από τον ευρωπαϊκό ένα αέριο χώρο. Δεν θα λειτουργούσε. Και θα καταλήγαμε ένα σύστημα το οποίο δεν θα μπορούσε να ενταχθεί σε ένα παγκόσμιο σύστημα, διότι ο εναέριος χώρος, το μεγαλύτερο ποσοστό του εναερίου χώρου του κόσμου είναι πάνω από τους ωκεανούς και δεν ανήκει σε κάποια χώρα. Άρα δεν θα λειτουργούσε αυτή η λύση. Τι κάναμε για να το αποφύγουμε αυτό. Ε, μια κινέζικη αεροπορική γραμμή, η αμερικανική γραμμή που πετάει, εταιρεία μάλλον που πετάει στην εταιρεία, πρέπει να υπόκειται στην ίδια αρχή του ορυπέρων πληρώνει, όπω και οι ευρωπαϊκέ αεροπορικέ εταιρείε που πάνε από την Ευρώπη και πάνε στην Ασία και πάνε στι Πολιτείε. Πρέπει να υπάρχει παράλληλη αντιμετώπιση. Αυτό ακριβώ κάνουμε. Να πω επίσης για τα αντίπεινα που φοβόσαστε. Φανταστείτε το εξή. Έχουμε ένα νόμο στην Ευρώπη που θεσπίστηκε πριν από τρία χρόνια. Πλησιάζει η ημερομηνία εφαρμογή και την ημέρα αυτή λένε οι Κινέζοι και αναφέρεται στους Financial Times στο πρωτοσέλιδο, όπως έγινε την Άνοιξη, ότι αν δεν αλλάξετε την νομοθεσία σας, τότε θα λάβουμε διάφορα μέτρα αντιπίνων και δεν θα παραγγείλουμε στην τάδε δίνα εταιρεία η Επιτροπή Βιομηχανίας των ΗΠΑ θα συμφωνεί. Εάν αρχίσουμε να υποχωρούμε επί τη βάση τέτοιων απειλών, η Ευρώπη θα βρεθεί σε πολύ δυσχερή θέση. Θα συμφωνεί και η Επιτροπή σας. Και δεν θα είναι ενδιαφέρον να είσαστε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να είστε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι κάθε φορά που κάποιο απειλεί την νομοθεσία μας θα την αλλάζουμε. Δεν είναι βιώσιμη λύση αυτή την Ευρώπη. Πιστεύω ότι οι Αμερικανοί έλυσαν ένα θέμα, ε, ε, ε, υπήρξε προσφυγή στα αμερικανικά δικαστήρια από τις εταιρείες, αεροπορικές εταιρείες. Δεν ξέρω θα κάνουν το αντίστοιχο και σε εμά. Η Φιώνα Χολ αναφέρθηκε για την έμεση αλλαγή της χρήσης των γεών και την ποιότητα των καυσίμων που σχετίζονται τα δύο. Δεν μπορώ να πω σε λεπτομέρειες για την πρότασή μας. Δεν τελείωσε η δουλειά, γι' αυτό δεν κάναμε την πρόταση. Είναι σημαντικό να υπάρχει ένας παράγων συντελεστής για την έμεση αλλαγή χρήσεως των γεών. Πρέπει να δεχτούμε ότι συμβαίνει αυτό. Και ότι έχει απεσυνέπειες. Βλέπουμε αλλαγή στην Αφρική εδάφη που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή τροφίμων στην Αφρική χρησιμοποιείται για φυτά που παράγουν καύσιμα για μας. Αυξάνεται η τιμή των τροφίμων και γι' αυτό συζητείται με σοβαρό το θέμα, γιατί θα έχουμε σοβαρά προβλήματα εάν ε, δεν το προσεγγίσουμε σωστά. Για το CDM να υπάρχουν προβλήματα Το αλλάζουμε ο 1η πρώτου 2013 το CDM στην Ευρώπη. Από πρώτου 2013 η Ευρώπη ήδη το καλύπτει το θέμα αυτό από την νομοθεσία. Ότι δεν θα έχουμε νέους μηχανισμούς καθαρής ανάπτυξης και σχετικά προγράμματα νόμιμα στις αναδυόμενες αλλά στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και στις ευάλωτες προβληματικές χώρες για να προωθήσουμε τα προγράμματα σχετικά. Και συνεργαζόμαστε με τον Επίτροπο Πίμπαλτς και όχι η κυρία Πίμπαλτς. Το θέμα αυτό δεν είναι προϋπόθεση για τη δεύτερη περίοδο αναρρίψης υποχρεώσεων. Έχουμε άλλους όρους. Ήδη αλλάξαμε τη δική μας νομοθεσία σχετικά με αυτό. Και μπορούμε να σταματήσουμε, Πρόεδρε. Είναι ξεκάθαρο, θαρό Ότι αν δίνουμε δισεκατομμύρια στην Ευρώπη και τα δίνουμε προς για να χρησιμοποιούν καλύτερες τεχνολογίες οι ανταγωνιστές μέσω του CDM χωρίς να συνεργαζόμαστε με τις αναπτυσσόμενες χώρες δεν θα πετύχουμε. Γι' αυτό αλλάξαμε και το χρονικό όριο των τριών ετών. Νομίζω ότι καλύπτω και το ερώτημα του κυρίου Ρόλτς. Θα συνεργαστούμε με τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και θα αλλάξουμε το CDM, τους μηχανισμούς αυτούς, σε μια χούφτα χωρών πήγαιναν 7% τα προγράμματα. Ινδία, Κίνα, Βραζιλία, Κορέα ήταν οι μεγαλύτεροι αποδέκτες των πόρων και των προγραμμάτων. Άρα είναι λογικό αυτό να αλλάξει. Το καταλαβαίνετε γιατί. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση αυτή, τις πληροφορίες, ε, την ευκαιρία να ανταλλάξουμε επιχειρήματα. Τώρα βλέπω η ώρα έχει τελειώσει γιατί και οι διερμηνείς έχουν δικαίωμα να κάνουν διάλειμμα. Α, δύο συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Η κυρία Μέρκης, σύντομα όμως σας παρακαλώ. Ναι, θέλω να ρωτήσω κάτι. Να κάνω κάποια σχόλια για την αεροπορία. Βεβαίω, σας στηρίζω πλήρως ε, όσον αφορά την, ε, το εμπόριο εκπομπών ε, και οι περισσότερες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείε δεν έχουν πρόβλημα, αλλά αν χάσουν τα δικαιώματά τους, να μπουν π.χ. στο ρωσικό εναέριο χώρο για να πάνε στην Ασία και μπορεί κάλλιστα ε, να τα χάσουν τα δικαιώματα αυτά, τότε χάνουν ε, το 1 τέταρτο του τζίρου τους. Ε, δεν γίνεται. Δεν είπα να αλλάξουμε το πρόγραμμά μας αλλά ίσως την, θέση ενισχύει. Να το καθυστερήσουμε λιγάκι. Για μήνες μιλάω έτσι, όχι χρόνια. Το καταλάβαμε όλοι το πρόβλημα νομίζω. Και δόθηκε μια απάντηση. Κυρία Κολάρσκα Μπομπίνσκα, στα διάφορα θέλω να πω κάτι. Θέλω να προσκαλέσετε τον Επίτροπο Έτιγκερ σε μια μελλοντική συνεδρίαση για να μας πει τα των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσία για την εφαρμογή του τρίτου πακέτου. Ευχαριστώ. Έξυπνη πρόταση. Να προσπαθήσουμε. Δεν είναι εύκολο να βρούμε ημερομηνίες με τους επιτρόπους. Σήμερα τα καταφέραμε. Οπότε σας ευχαριστώ. Ή και η κυρία Χέντεγκαρτ βεβαίως μπορεί να απαντήσει για να το ξέρετε, ε, αυτό το μήνα θα έρθουν εμπειρογνώμονε από τη Ρωσία στι Βρυξέλλες για να συζητήσουν με του δικού μα. Εγώ πήγα και στη Μόσχα την προηγούμενη εβδομάδα και το συζήτησα μεταξύ πολλών άλλων. Να το ξέρετε, δεν είναι ότι καθόμαστε και περιμένουμε τι θα γίνει. Και κάτι ακόμα. Ναι, πρώτη πρώτου 2012 τίθεται νομοθεσία, αλλά ήδη τους είπαν η κάθε νομοθεσία, πόσες δωρεάν άδειε θα έχουν, έχουν πολλές δωρεάν άδειε. οπότε μέχρι το 2013, δηλαδή έτσι είναι ο νόμος, θα τους επιστρέψουν τα λεφτά και τα λοιπά. Οπότε έχουμε χρόνο. Ε, δηλαδή μην σκέφτεστε ότι είναι 10 Νοεμβρίου και 1 Ιανουαρίου θα ισχύσει. Όχι, έχουμε όλο το 2012.